Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας και θα μιλήσω αν μου επιτρέπετε στη γλώσσα μου. Θα μιλήσω εν μέρη ε, στα τσέχικα και εν μέρη στα αγγλικά. Καλημέρα σας. Ε, συνεχίζεται λοιπόν η συνεδρίασή μας και ας συνεχίσουμε ε, με το σημείο υπαριθμών 7 που είναι η σύσταση για τη ε, δημιουργία της, ε, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης. Η συγητής είναι η κυρία Βόλτμαν η οποία έχει και το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα και εγώ να μιλήσω σήμερα το πρωί στη μητρική μου γλώσσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω αναφέροντα σήμερα το πρωί ότι είμαι ιδιαίτερα... Α, να σας περιμένω μια στιγμή. Δηλώνω λοιπόν με μεγάλη ικανοποίηση ε, για το γεγονό ότι έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προπολογισμό για την αύξηση τη εξωτερική παρέμβαση κατά 30%. Από τα 94,5% ε, εκατομμύρια μάλλον στα 122 εκατομμύρια για την περίοδο 2021-2027. Και επέλεξε έναν πιο απλό και πιο ευέλικτο προπολογισμό και τα δύο είναι πολύ ε, απαραίτητα. Πέραν τούτου, η εκπρόσωπος, εκπρόσωπο, με την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προέτεινε και ένα νέο μηχανισμό πέραν του προπολογισμού, το οποίο θα εξετάσουμε σήμερα. Τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ασφάλεια. Με 10,5 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη πραγματική περίοδο. Πέρυσι ε, συμφωνήσαμε με την ε, ε, το μηχανισμό υποστήριξης ε, της ανάπτυξης και μια συμβολή στον μηχανισμό ειρήνης, κάτι το οποίο ε, επιτρέπει την παροχή στρατιωτικής βοήθειας και αερογής σε τρίτες χώρες. Θα προαγάγει λοιπόν αυτός ο μηχανισμός την ασφάλεια και τα σταθερότητα και την ειρήνη με τη χρηματοδότηση διαφόρων στρατιωτικών χωρίς ε, να συνδέεται με αυστηρούς ε, κανόνες και προϋποθέσεις ε, ανάπτυξης. Σε ορισμένες χώρες αυτή η βοήθεια μπορεί να είναι πολύ σημαντική. Σκεφτείτε τις χώρες όπου λόγω έλλειψης ασφάλειας δεν μπορούμε να έχουμε πολιτικούς φορείς. Γι' αυτό θα πρέπει να προστατεύσουμε τις στρατιωτικές μας, τους στρατιωτικούς μας πόρους δεν ξέρω κατά πόσο τώρα θα ε, άρουμε τυχόν περιορισμούς και δυσκολίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα η στήριξη αυτή χρηματοδοτούνταν μόνο αμέσω του μηχανισμού Ατένα. Και περιοριζόμασταν μόνο σε επιχειρήσεις υπό αφρικανική ηγεσία μέσω του μηχανισμού για την Αφρική. Τώρα με αυτό τον μηχανισμό αυτό θα αλλάξει. Ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ασφάλειας λοιπόν θα τα αλλάξει όλα αυτά. Θα καλύψει το κοινό κόστος των ε, επιχειρήσεων σε σχέση με το μηχανισμό Αθήνα. Έτσι τα κράτη-μέλη πιο γρήγορα θα μπορούν ε, και θα παροτείνονται να συμμετέχουν σε ορισμένε επιχειρήσει. Σε δεύτερον, θα καλύπτει και επιχειρήσει Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζοντα τι τρίτε χώρε όχι μόνο στην Αφρική αλλά και πέραν αυτής. Τρίτον, θα καλύψει και δραστηριότητες ε, σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση δυναμικού ε, στο στρατιωτικό επίπεδο, κάτι το οποίο εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό, κατάρτιση, υποδομές, ε, εξοπλισμό, και έτσι είμαι πεπισμένη ότι αυτός ο νέος μηχανισμός θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα ε, των επιχειρήσεών μας, γιατί τώρα κάποιες φορές κάνουμε εκπαιδεύσει και καταρτήσεις, αλλά είναι αναποτελεσματικές, γιατί οι εταίροι μας ε, δεν έχουν επαρκείς ικανότητες. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Ασφάλειας, Ειρήνη, συγγνώμη, θα επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενδυναμώσει τους εταίρους τη και να τους βοηθήσει βοηθήσει για να διαχειριστούν καλύτερα τις κρίσεις, να αποτρέψουν ε, συγκρούσεις και να ε, διασφαλίσουν τη σταθερότητα. Και η σταθερότητα των εταίρων μας ε, είναι πολύ σημαντική για εμάς και προς το συμφέρον μας. Όπως γνωρίζετε, οι δραστηριότητες με προεκτάσεις στον στρατιωτικό τομέα δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό βάσει του άρθρου 24.2. Γι' αυτό και δημιουργείται αυτό το νέο εργαλείο. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ειρηνή, ε, λοιπόν, θα χρηματοδοτηθεί ε, με χρηματοδότηση και των κρατών μελών, με βάση κλίδα κατανομής, ε, βάσει του ακαθάριστου εθνικού προϊόντο. Έχουν υποβληθεί προτάσεις για ενέργειες, μετά το Συμβούλιο ε, Άμυνας Ομοφόνος αποφασίζει για τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν. Όπως κάθε άλλο χρηματοδοτικό μέσο, η υλοποίηση και εκτέλεση δηλαδή, του προπληγισμού ε, θα εναπόκειται στην ύπατη εκπρόσωπο με στήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. και ε, αρμόδια ε, μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αναλάβει και την υλοποίηση καθώς και από την ε, αντίστοιχη επιτροπή και με εκπροσώπους των πρώτων μελών και με εκπρόσωπο της ΥΠΑ της εκπροσώπου. Από τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία εγώ θα ήθελα να σταθώ. Πρώτον, οι λόγοι για τους οποίους χρειαζόμαστε αυτό το μηχανισμό. Γιατί θα συμπληρώσει τυχόν κενά που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χρηματοδότησή μας. Είναι ευέλικτος μηχανισμός και θα επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ταχύτερα και πιο συχνά να παρεμβαίνει όταν υπάρχουν κρίσεις, ε, όταν μας το ζητάνουν οι εταίροι μας ή όταν εμείς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη μία τέτοια συνεισφορά. Δεύτερον, κάτι που για το Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει επαρκής δημοκρατικός έλεγχος από το Κοινοβούλιο το οποίο θα πρέπει να ε, ενημερώνεται εγκαίρως και πλήρως και να υπάρχει μάλιστα και διαβούλευση με αυτό πριν τη λήψη αποφάσεων. Και τρίτον, ε, ζητούμε το Συμβούλιο να μας διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν ενέργειες που θα αντιβαίνουν ε, στο διεθνές δίκαιο. Εν γέννη, θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι να τον πιο ευέλικτος, γιατί εκεί έγκυται και η προσθέμενη αξία για εμάς. Το Συμβούλιο Ε, μπορεί να μην δίνει ε, επαρκή χώρο στο Κοινοβούλιο για τον προπολογισμό αυτών. Γι' αυτό εμεί όμω ζητούμε το αντίθετο. Περιμένω τι τροπολογίε σα μέχρι τι 24, συγγνώμη, 4 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Βόλτμαντς ε, για την παρέμβασή σας. Πριν λοιπόν ξεκινήσει η συζήτηση, έχω μία ερώτηση προς εσάς κυρία Βόλτμαν. Αν κατάλαβα καλά, μιλήσατε για συνεισφορές ε, με βάση το GNI, αλλά εγώ δεν έχω πολύ καλή εμπειρία με αυτές τις ε, συνεισφορές της GNI Τι ε, συνεισφορέ με βάση το ΑΕΠ μάλλον, το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, στον προπολογισμό του ΝΑΤΟ. Ε, γι' αυτό λοιπόν δεν ξέρω, ε, τα κράτη-μέλη θα το δεχτούν αυτό, δηλαδή η συνεισφορά του να βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα. Ο κύριος Γκάλα έχει το λόγο, παρακαλώ. Είναι σκιώδης εισηγητής. κύριος ε, Ντανζόν είναι σκιωτισηγητής, αλλά δεν είναι παρόν και ζήτησε από εμένα να ε, παρουσιάσω τη δική τη θέση. Λυπάται πάρα πολύ που δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα το πρωί. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για την έκθεσή της και στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να συστήσει το των δυνατόν αυτό το νέο εργαλείο, τη διευκόλυνση ή το μηχανισμό για την ειρήνη. Πρόκειται για έναν νέο προϋπολογισμό 10,5 δις για 7 χρόνια, ένα νέο ταμείο και θα καλύπτει μόνο εκείνες τις δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω περιπλοκών που ενδεχομένω να υπάρξουν στον αμυντικό τομέα και όλα αυτά σε απόλυτη συμφωνία με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός λοιπόν ο μηχανισμός θα χρηματοδοτεί ε, τις κλασικές δαπάνες των ε, στρατιωτικών επιχειρήσεων και έτσι θα αντικαταστήσει το μηχανισμό Αθήνα. Επίσης ε, θα συμβάλλει και σε άλλες επιχειρήσεις, στρατιωτικές, υποστήριξης όμως επιχειρήσεις που διεξάγουν άλλοι παράγοντες, ξένοι και έτσι θα αντικαταστήσει τον Αφρικανικό Μηχανισμό ε, Στήριξης για την ειρήνη, θα συμβάλλει στην ειρήνη, πρόληψη ε, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη και ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας. Όλα αυτά εντάσσονται και μέσα σε αυτό που ήδη έχουμε στην ε, δημιουργία ικανοτήτων για την ειρήνη και την ανάπτυξη. Αυτά λοιπόν θα επιτρέψουν να χρηματοδοτείται ένα μεγαλύτερο ποσοστό του κλασικού κόστους ε, για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο στόχος αυτού του νέου εργαλείου βεβαίως ε, και είναι ευπρόσδεκτος και ο στόχος είναι και πολύ φιλόδοξος, είναι όμως και περίπλοκος και πάρα πολύ τεχνικός, κυρίως σε θεσμικό επίπεδο. Απομένουν πολλές αναπάντητες ερωτήσεις όπω όπως η δομή του μηχανισμού, το πώς θα, το διαχειρίζεται, πώ θα διοικείται και ο ρόλος των κρατών μελών. Επίσης η αύξηση των κλασικών δαπανών δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη μείωση οποιαδήποτε μείωση των υποχρεώσεων. Ο ε, κ. Ντανζόν προσβλέπει στην αγαστή συνεργασία με τον εισηγητή και με τους, ε, την εισηγήτρια μάλλον και τους εισηγητές για αυτή την έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκάλερ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Φραντζούλικα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της και θέλω να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια κάναμε κάποια βήματα προς τα Εμπρό στον τομέα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας. Και κατευθυνόμεθα προς ένα πολύ σημαντικό στόχο που είναι η σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άμυνας. Όσον αφορά τώρα τόσο το δυσκολότερο διεθνές περιβάλλον και τη μεγάλη σημασία που αποδίδουν οι πολίτες μας στην ασφάλεια, θα ήθελα να πω ότι οι Ευρωπαϊκή εταίροι περιμένουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στη δική μας την περιοχή, αλλά και πέρα από αυτήν. Με αυτή την έννοια πρέπει να ενισχύσουμε τις πράξεις μας για να ε, προβλέπουμε τις ε, συγκρούσεις και εγώ χαιρετίζω την πρόταση να συσταθεί αυτός ο μηχανισμός και αναγνωρίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα εργαλείο έτσι ώστε ε, να βελτιωθεί η ικανότητα των εταίρων μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να επιλύσουμε ορισμένα σημαντικά προβλήματα του ευρωπαϊκού αρχιτεκτονήματος για τη χρηματοδότηση τη Ειρήνη και τη ανάπτυξη με βάση ε, τις δικές μας τις αλλά και λεπτομερή ανάλυση των αναγκών των εταίρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα βασικά στοιχεία έτσι ώστε ο μηχανισμό αυτό να μπορεί να καλύπτει το στόχο του για την διατήρηση τη ειρήνη. Πρώτον, να υπάρχει ένα μηχανισμό έτσι ώστε να υπάρχει ουσιαστική γενική εικόνα τόσο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιμένω επ' αυτού η ενίσχυση είναι καθοριστικό ρόλο, αλλά και αρμοδιότητες σε επίπεδο εθνικών κρατών μελών που χρηματοδοτούν αυτό τον μηχανισμό. Δεύτερον, όσον αφορά την βελτίωση των ικανοτήτων, Εδώ υπάρχει έλλειψη ασφάλειας στην Αφρική. Αυτό θέλω να επισημάνω. Και αυτό οφείλεται κυρίω στα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τον μηχανισμό ειρήνη στην Αφρική. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Ειρήνης είναι απαραίτητος έτσι ώστε να προσφέρεται σταθερή προβλέψιμη χρηματοδότηση στις ε, πρωτοβουλίες της Αφρικανικής Ένωσης για την ειρήνη και στις σχετικές αποστολές. Αυτός ο νέος μηχανισμός θα αντικαταστήσει τον μηχανισμό της Αφρικής και τον μηχανισμό Αθήνα με στόχο να αρθούν τα εμπόδια και επίση στόχο να διευρυνθεί ε, το πλαίσιο των κλασικών δαπανών που θα χρηματοδοτούνται. Εγώ ε, συμφωνώ ότι πρέπει να πλουστευτεί ο μηχανισμός για να χρηματοδοτούνται οι αποστολές της ε, κοινή πολιτικής άμυνας και ανάπτυξης. Επίσης, πρέπει να γίνονται σεβαστές οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ανθρωπιστικά θέματα. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι πρέπει να υπάρχουν βέβαια και απαραίτητοι μηχανισμοί. Με την η διαχείριση αυτού του εργαλείου, του μηχανισμού είναι πολύ σημαντική αν μας ενδιαφέρει να επιτευχθεί ο στόχος που είναι να στηριχθούν οι ε, χώρες για να προσφέρουν μια ασφαλή βάση έτσι ώστε να υπάρχει οικονομική και πολιτική ε, βιωσιμότητα με βάση τους στόχους που έχουν καθαριστεί. Τέλος, ο μηχανισμός αυτός πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες φιλοδοξίες για την ασφάλεια και την άμυνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Φραντζούλικα, λέω πρόεδρος, και πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ μαζί σας αλλά συμφωνώ και με τον κύριο Ντανζά ή τον κύριο Γκάλερ ότι πράγματι αυτό το εργαλείο είναι πολύ σημαντικό. Αλλά όπως όλοι μας γνωρίζουμε, ε, τα καλά πράγματα είναι χρονοβόρα και μερικές φορές η όλη διαδικασία είναι επώδυνη. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να φάσουμε στη φάση όπου θα έχουμε ένα αποτελεσματικό μηχανισμό. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Πρέπει βέβαια ευθύ εξ αρχή να πω ότι η δική μου η πολιτική ομάδα αυτόν τον μηχανισμό τον αντιμετωπίζει πολύ επιφυλακτικά. Ε, σχεδόν και τον απορρίπτουμε, θα τολμούσα να πω. Θεωρούμε ότι η λέξη, ε, ο τίτλος ε, «Μηχανισμός διατήρησης ειρήνης» είναι παραπλανητικός. Εδώ, κατ' ουσίαν, πρόκειται για ένα αμυγός στρατιωτικό εργαλείο. Όσον αφορά τώρα την τεχνική η εφαρμογή του όλου θέματος, θέλω να πω, ε, έχει αναφερθεί και υποστηριχθεί ότι κατά το παρελθόν υπήρχαν δυσκολίες να διεξάγονται επιχειρήσεις ή να χρηματοδοτούνται αμυντικά μέτρα. Και πολύ σωστά γίνεται επισήμανση στο άρθρο 41.2 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο μηχανισμός ειρήνης, ε, γι' αυτό το λόγο ε, τοποθετείται εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θέλω να σας πω ότι στηρίζω το αίτημα που είναι σωστό σχετικά με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν υπάρχει άμεσος έλεγχος αυτού του εργαλείου, γιατί αυτό το εργαλείο εντάσσεται εκτός του, ε, του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηρίζουμε αυτό που είναι στο εδάφιο R και στο 1αβ ABCDE, ε, επίσης το 2D, αυτά τα σημεία τα στηρίζουμε. Ε, όσον αφορά τώρα τις διαβουλεύσεις και την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκεί θέλω να σας πω, έχουμε μία μακρά εμπειρία και Μέχρι τώρα δυστυχώς δεν μπορούσε να υπάρξει αποτελεσματικός κοινοβουλευτικός έλεγχος και φοβάμαι ότι αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλλον. Κάτι άλλο στην έκθεσή σας πρόκειται για την διασύνδεση ασφάλειας και ανάπτυξης. Ο στρατός σε αυτό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, μα και βεβαίως και εγώ πιστεύω ότι η ασφάλεια και η ανάπτυξη μάλλον να το πω αλλιώς, ότι η ασφάλεια προϋποθέτει την ανάπτυξη. Το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να επιτύχει αυτήν την ασφάλεια. Ο προλαλής σας ε, μίλησε για το ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια προληπτική προσέγγιση και ανέφερε ότι θα πρέπει να υφίσταται ε, μια βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη. Ε, μίλησε και για τα κοινωνικά ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι όλα αυτά μπορούμε να τα επιτύχουμε με πρόληψη και με στρατιωτική εκπαίδευση, ούτε και με εξαγωγή όπλων, αλλά ούτε και με ε, συνεργασία ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο αυτών των αποστολών ειρήνης. Εξάλλου έχουμε και σχετική εμπειρία. Για δέστε τι έγινε με το Κονγκό, τη Σομαλία, το Αφγανιστάν, το Μαλί. Ε, υπάρχει μία κλιμάκωση στις εξαγωγές όπλων και εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι λυπηρά γεγονότα και δυσάρεστη εμπειρία. Αν λοιπόν πραγματικά θέλουμε ε, ένα σταθερό περιβάλλον, βιώσιμο περιβάλλον, τότε μόνο η κοινωνική βιωσιμότητα μπορεί να αποτελεί εχέγγυο. Οτιδήποτε άλλο απλά είναι πρόφαση για να υπάρχει πρόσβαση στους ε, πλουτοπαραγωγικούς πόρους και όχι για να αντιμετωπιστεί η ακραία φτώχεια. Πάρα πολλοί οργανισμοί έχουν καταστήσει σαφές ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει πάντα να είναι ουδέτερη και ως εκ τούτου ανεξάρτητη από παρεμβάσεις ε, στρατιωτικές. Η μη στρατιωτική συνεργασία είναι εκείνη, όπως αναφέρεται εδώ, η οποία καταστρέφει την ουδετερότητα και θέτει και σε κίνδυνο τους ε, συνεργάτες των ανθρωπιστικών προγραμμάτων. Αυτό έχει καταστεί σαφές επανειλημμένα. Και τέλος, θέλω να πω ότι το εργαλείο αυτό δεν είναι προσαρμοσμένο ε, στο να αντιμετωπίζει κρίσεις, αλλά κατ' ουσίαν είναι ένα κρυφό εργαλείο για τη μετανάστευση για την παρεμπόδιση μετακίνηση μεταναστών. Και είναι ένα εργαλείο για στρατιωτικά και όχι για μη στρατιωτικά μέτρα. Τέλο, όσον αφορά το μηχανισμό ειρήνη που υποτίθεται θα αντικαταστήσει το μηχανισμό Αθηνά και να τον διευρύνει, θέλω να επισημάνω ότι στο μέλλον όλα τα κράτη-μέλη τα οποία καταβάλουν συνδρομή σε αυτό το μηχανισμό αυτόματα συμμετέχουν και ε, σε όλες τις άλλες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαγωγή όπλων και πάρα πολλά άλλα. Ακόμα και αν το ίδιο το κράτος μέλος δεν δραστηριοποιείται, δηλαδή δεν διαθέτει ένοπλες δυνάμεις. Εδώ ισχύει αρχή «Coast lie where they fall», η οποία πλέον ακυρώνεται. Εγώ θεωρώ ότι ορισμένες ε, χώρες, εντάξει αυτό βρίσκω θετικό πρέπει να πω, ε, ότι ορισμένες ε, χώρες θα καταφύγουν στην ρήτρα εξαίρεσης. Και αυτό το βρίσκω καλό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Είπατε, κυρία μου, ότι γίνεται λόγος για τη χρηματοδότηση ενός στρατιωτικού μέσου και αυτό δεν αντιστοιχεί στους στόχους. Δεν πρόκειται περί αυτού, πρόκειται περί της ειρήνης. Κυρία Λέζιγκε, πρέπει να σας πω ότι ως δημοσιογράφος είχα εργαστεί στις ε, ζώνες, στις εμπόλεμες ζώνες όπου υπήρχαν σειράξεις και έχω δει με τα μάτια μου ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη εάν δεν καταπολεμήσουμε τη βία. Επομένως αυτό το μέσο που έχει να κάνει με τη στρατιωτική χρηματοδότηση μπορεί να πετύχει τους σκοπούς και να εφέρει την ειρήνη. Ο κύριος Γιούρεκ είναι επίσης σκιώδης εισηγητής. Θέλετε να παρέμβετε με αυτή σας την ιδιότητα ή όχι. Εάν όχι, πολύ καλά. Έρχομαι τώρα στον κύριο Γκάλερ που θα ήθελε να πάρει το λόγο ξανά. Παρακαλώ κύριε Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα δεν ε, ομιλώ εξ ονόματος του κυρίου Ντονζό, του σκιώδη ηγητού, αλλά θα ήθελα εγώ να τοποθετηθώ κάπως γενικά. Κοιτάξτε, για πάρα πολλά χρόνια στην υποεπιτροπή μας συζητήσαμε για το πώς είναι δυνατόν να μεταρρυθμίσουμε αυτόν τον μηχανισμό ε, Αθήνα δηλαδή πώς μπορούμε να περιορίσουμε ε, τις ε, κοινέ δαπάνες ε, κατά 10% περιορισμός των γενικών δαπανών και αυτό το είχαμε προτείνει για ένα καθαρά ρεαλιστικό λόγο. Δηλαδή, στην πράξη συμβαίνει. Οι δαπάνε για στρατιωτικέ επιχειρήσει δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δεν αλλάξουν, δεν τροποποιηθούν οι συνθήκε, δεν θα αλλάξει και αυτό. Αποτέλεσμα, αυτό το ξεχωριστό ταμείο που το λέγαμε Αθήνα, γι' αυτό το λόγο συστήθηκε, για να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Κατ' ουσίαν πρόκειται για την κοινή χρηματοδότηση, παραδείγματο χάρη, Ε, των ε, ε, κεντρικών εγκαταστάσεων για μια επιχείρηση, δηλαδή όχι χρηματοδότηση συσκευών, εξοπλισμών και οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είχε ως συνέπεια το εξής. Οι χώρες οι οποίες παρότι είχαν συμφωνήσει επί της ουσίας, δεν είχαν όμως την οικονομική δυνατότητα να καλύπτουν οικονομικά το προσωπικό τους, αυτές ε, απήχαν με αποτέλεσμα εκείνοι οι οποίοι είχαν κάποια οικονομική δυνατότητα, ήταν εκείνοι οι οποίοι κατά κύριο λόγο έπρεπε και καλούντο να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι είναι πιο ε, δίκαιο, εφόσον αποφασίζουμε όλοι από κοινού για μια πολιτική, τότε να επιμεριζόμαστε και τις δαπάνες. Αποτέλεσμα, ας πούμε, σε αποστολές, που, σε επιχειρήσεις θαλάσσιας μορφής. Υπάρχουν χώρες και η συνάδελφος κυρία Γκόμες αναφέρει συνεχώς ε, τη δική συμπατρίδα. Η Πορτογαλία έχει ένα σχετικά μεγάλο στόλο ε, και οι Έλληνες, αλλά δεν έχουν οικονομική δυνατότητα. Αποτέλεσμα λένε εμείς δεν θα συμμετέχουμε και θα παραμείνουμε εκεί που είμαστε. Τώρα, αν μπορούσαμε να επεκτείνουμε, όπως σα είπα, τον επιμερισμό των δαπανών, ίσως θα μπορούσαν να συμμετέχουν περισσότερο και η Πορτογαλία και η Ελλάδα με αποτέλεσμα, ε, λογικό επακόλουθο, οι άλλοι που συμμετέχουν περισσότερο να αποσυρθούν λιγάκι και το λέω επανειλημμένα και στη Γερμανία. Έχω την εντύπωση ότι το Υπουργείο Οικονομικών το κατάλαβε, αλλά κάποια άλλα Υπουργεία δεν το έχουν κατανοήσει. Και λέω λοιπόν, εάν ε, μπορούμε να μη συμμετέχουμε έστω και καταβάλλοντας κάποιο ποσό, τότε νομίζω ότι αυτό θα ήταν μία συνεισφορά και μία εξέλιξη για μας που θα μας οδηγούσε στο να μην κάνουμε υπερβολικές ε, σπατάλες και δαπάνες. Με λίγα λόγια, αυτός ο μηχανισμός ε, ειρήνης κατά την άποψή μου, επιμερίζει καλύτερα το βάρος. Στο, σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών έχουμε χώρες οι οποίες ε, ε, χρηματοδοτούν ε, τις στρατούς τους ή συνεισφέρουν, ξέρετε πώς, μόνο με το που σηκώνουν το χέρι. Το Νεπάλ, η Σρι Λάγκα, αυτές οι χώρες δεν θα μπορούσαν καν να έχουν στρατό αν δεν συμμετείχαν σε επιχειρήσεις ε, υπό την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών. Κατόπιν τούτου θεωρώ ότι θα πρέπει πράγματι να συμμετέχουν και αυτές οι χώρες, να επιμεριζεί το κόστος. Έτσι θα υπάρχει και καλύτερη συντήρηση των εξοπλισμών και καλύτερος επιμερισμός του βάρους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Γκάλερ. Θα ήθελα να ξέρω. Θέλει κάποιος άλλο το λόγο. Εάν όχι... Στρέφομαι προς την εισηγήτρια για να απαντήσει στις ερωτήσεις και στα σχόλια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο ερώτημα βεβαίως που θέσατε εσεί. Θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη θα συμμετάσχουν σε αυτό το σύστημα γιατί με αυτό το σύστημα θα καλύπτεται μεγαλύτερο κομμάτι των, κοινών δαπανών. Από το 10-15% πάμε στο 30-35%. Επομένω, θεωρούμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να πείσουμε και τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν στο σύστημα. Πρέπει να πω ότι γενικά άκουσα θετικές παρατηρήσεις για την αναγκαιότητα θέσπισης αυτού του μηχανισμού, την ευελιξία του, ε, ότι υπάρχει πλέον μεταρρύθμιση ε, και επανεξέταση του ε, Ατένα, που ήταν κάτι το οποίο θέλαμε εδώ και πολλά χρόνια. Για αυτά που είπε η κυρία Λόζινγκ, από τη δική σου πολιτική ομάδα, βέβαια, για να είμαι ειλικρινή, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Περίμενα να είστε επικριτικοί απέναντι σε αυτή την πρόταση, είστε γνωστοί γι' αυτό στο Κοινοβούλιο. Να πω με κάθε ειλικρίνεια ότι η ασφάλεια, η ανάπτυξη και οι στρατιωτικέ επιχειρήσει πάνε χέρι-χέρι και πρέπει να τολμήσουμε να επενδύσουμε και για την ανάπτυξη ε, ικανοτήτων. Συμφωνώ για την ε, εποπτεία από το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι τα πήγαμε πολύ καλά σε αυτό και το επισημάνομαι σαφώ, αλλά περιμένω φυσικά με ενδιαφέρον τις τροπολογίες τις οποίες θα εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση για αυτό το θέμα. Θα ήθελα μόνο να σας υπενθυμίσω ότι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 4η Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Στη συνέχεια στις 21 και στις 22 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε το κείμενο στην Επιτροπή μας και θα συζητηθεί το κείμενο στην Ολομέλεια του Μαρτίου του 2019. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Λέσιγκερ. Μπορούμε να αλλάξουμε. Μπορείτε να έρθετε εδώ στο Προεδρείο να προεδρεύσετε. Γιατί θα έχουμε ακρόαση στη συνέχεια. Παρακαλώ. No, no, no. I have to go because I have another program. Ja, Καλημέρα σας. Λοιπόν, και πάλι καλημέρα σας και θα ήθελα να καλωσορίσω κυρίως τους εμπειρογνώμονές μας. Ε, ελπίζω το γεγονός ότι ξεκινάμε λίγο νωρίτερα, βέβαια πρόκειται για ακρόαση, ελπίζω να μην είναι αυτός ο λόγος που δεν ε, έχουμε ακροατήριο, ικανοποιητικό ακροατήριο. Σήμερα θα μιλήσουμε για την χρήση των τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε συζητήσει αρκετά συχνά για το θέμα αυτό και στην Επιτροπή μας και μάλιστα έχουμε συντάξει και ένα σχετικό ψήφισμα. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να μου επιτρέψετε ε, τις δικές μου τις προσωπικές απόψεις να τις καταθέσω αργότερα θα τις ε, καταθέσω με τη μορφή ερωτήσεων και αυτές τις ερωτήσεις θα τις ε, καταθέσω όχι τόσο με την ιδιότητά μου της Προέδρου αλλά μετά από εντολή της ε, πολιτικής μου ομάδας. Να καλωσορίσω τον στρατηγό Μισελ, γενικός γραμματέας για θέματα ασφάλειας στη Γαλλία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ε, εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Μπορώ να μιλήσω γαλλικά. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως είναι κάπως πιο εύκολο για μένα να μιλήσω γαλλικά. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και που μου δίνετε την ευκαιρία να παραστώ εδώ και να σας κάνω μια παρουσίαση για τον τρόπο με τον οποίο η γαλλική κυβέρνηση θέλησε εδώ και τέσσερα χρόνια να εργαστεί στον τομέα καταπολέμησης ε, των μη επανδρομένων αεροσκαφών, κυρίως των απειλών που προέρχονται από αυτόν και όχι των μη επανδρομένων αεροσκαφών αυτών καθεαυτών. Έχω κάποιες διαφάνειες στα αγγλικά για να παρακολουθήσετε τους βασικούς λόγους ε, για τους οποίους ξεκίνησε αυτή η δουλειά ε, και τα βασικά στοιχεία τα οποία έχουμε υιοθετήσει. Μιλούμε για μη επανδρομένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για κακούς σκοπούς, δεν έχει επιληθεί το πρόβλημα. Είναι ένα σύστημα, το σύστημα των drone, το οποίο εξελίσσεται, πολύ γρήγορα από τεχνολογική σκοπιά. Έχουν όλο και περισσότερες δυνατότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τρομοκρατικούς ή άλλους ε, ε, κακούς σκοπούς. Στη Γαλλία έχουμε καταγράψει τα τελευταία τέσσερα χρόνια 400 πτήσεις μη επεδρομένων αεροσκαφών σε επικίνδυνα σημεία και περιοχές συχνά οι νυχτοφύλακες, οι αστυνομικοί που περιπολούν τη νύχτα τον μπερδεύουν. Τον μπερδεύουν το μη επανδρομένο αεροσκάφο, το drone, με ένα ε, κανονικό αεροσκάφο πτήσης. Εν πάση περιπτώσει γνωρίζουμε ότι περίπου 300 τέτοιου είδους drone έχουν πετάξει πάνω από επικίνδυνα ή ευαίσθητα σημεία στην εθνική μας επικράτεια. Αυτό είναι ένα γεγονός. Επίσης έχουν υπάρξει συγκρούσεις μεταξύ ε, ντρόουν και αεροσκαφών. Βλέπετε την φωτογραφία στη διαφάνεια. Στο αεροδρόμιο του Κεμπέκ έχει συμβεί αυτό. Και αυτή την εβδομάδα από ανοιχτές πηγές μάθαμε ότι ε, ένα ε, αυστριακό ελικόπτερο έχει συγκρουστεί με ένα ντρόουν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Πάλι δεν υπήρξε καμία βλάβη και καμία ζημιά και κανένας τραυματισμός. Σε κάθε περίπτωση είχαμε περισσότερες από μία ε, των ε, εναέριων χώρων πάνω από πυρηνικά μας εργοστάσια. Γνωρίζετε ότι η Greenpeace πέταξε ένα ντρόν πάνω από ένα ε, πυρηνικό εργοστάσιο και ε, το κατέβασε πάνω στο πυρηνικό αντιδραστήρα με ένα ε, Σούπερμαν, με ένα κουκλάκι Σούπερμαν, ακριβώς για να αποδείξει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της Γαλλίας δεν είναι ε, απόλυτα θωρακισμένες και σφραγισμένες. Έχουμε επίσης συγκεκριμένες πράξεις κακόβουλες που έγιναν στη Βενεζουέλα το καλοκαίρι δύο ντρόουν μπροστά από τον πρόεδρο Μαδούρο πέταξαν με σκοπό να ανατιναχθούν, είχαν προγραμματιστεί όχι, για να προκαλέσουν τραυματίες στο προεδρικό θεωρείο και τα μέτρα που είχαν υιοθετήσει οι αστυνομικές αρχές της Βενεζουέλας επέτρεψαν να υπάρξει απόκρουση αυτών των ντρόουν και να τελικά να εκραγούν και να πυροδοτηθεί ο μηχανισμός έκρηξής τους που είχε προγραμματιστεί αλλού και όχι μπροστά στο προεδρικό θεωρείο. Και σε μια επίθεση καρτέλ στο Μεξικό είχαμε δύο χειροβοβίδες με ντρόουν πάλι που είχαν ρηφθεί και ε, στο, στη Συρία επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί ντρόουν κατά ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων drone που ήταν εξοπλισμένα με οβίδες, τα οποία ε, σύμφωνα με ρωσικές πηγές πληροφοριών πλοηγήθηκαν δεκάδες χιλιόμετρα κουβαλώντας αυτές τις οβίδες, τις οποίες έριξαν ταυτόχρονα σε δύο συγκεκριμένες ε, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σε δύο σημεία, με συνδυασμένο τρόπο. Τα ντρόν λοιπόν ναι είναι ένα παιχνίδι, ναι είναι ένας μοχλός οικονομικής ανάπτυξης εξαιρετικά σημαντικός και εξαιρετικά επίκαιρος, όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κακόβουλο τρόπο και αυτή η κακόβουλη χρήση μπορεί να προκαλέσει πολύ, πολύ αρνητικά αποτελέσματα και φαίνεται αυτό από τα παραδείγματα που σας παρουσίασε. Με αυτές τις διαπιστώσεις λοιπόν η γαλλική κυβέρνηση διάλεξε να, και επέλεξε να δουλέψει με την εξή λογική. Να διατηρήσει αυτό τον οικονομικό κλάδο και για τη γαλλική οικονομία και για την ευρωπαϊκή οικονομία, να πλαισιώσει τη χρήση των ε, ε, μη επανδρομένων αεροσκαφών εμπορικής και αστικής χρήσης και όχι στρατιωτικής και να πλαισιώσει αυτή τη χρήση με συγκεκριμένη νομοθεσία. Άρα ανάπτυξη με κανόνες και με ρύθμιση της αγοράς βάσει νομοθεσίας. Πρέπει να εργαστούμε και πάνω στο πεδίο της ασφάλειας για την ασφάλεια των ευαίσθητων εγκαταστάσεων και την ε, ασφάλεια του πληθυσμού. Συνδυάσαμε λοιπόν τις δύο προσεγγίσεις ως επίσημη γαλλική κυβερνητική πολιτική. Στον τρόπο δράσης μας λοιπόν προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο πρόληψης, εκπαίδευσης, αποτροπής και τελικά παράβασης και κύρωσης ε, ε, όλων αυτών που χρησιμοποιούν τα ντρόουν, τα μη επαδρομένα αεροσκάφη, με κακόβουλο σκοπό. Το πνεύμα λοιπόν της εργασίας μας είναι το εξής και το βλέπετε στην οθόνη. Από όλα τα ντρόν που πετούν, από όλο αυτό το νεφέλωμα, το σύννεφο των μη επανδρομένων αεροσκαφών, θελήσαμε να ταυτοποιήσουμε ποια συνεργάζονται, ποια σέβονται και τηρούν την εθνική νομοθεσία προς το παρόν. Άπαξ και τα προσδιορίσαμε αυτά. Επόμενο βήμα ήταν οι δυνάμεις ασφαλείας και τάξης να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στα ντρόουν που μας δημιουργούν ε, αμφιβολίες, που δεν ξέρουμε κατά πόσο τηρούν τους κανόνες και στα ντρόουν δηλαδή που πρέπει να ερευνήσουμε ε, περαιτέρω. Και άπαξ και γίνει αυτή τη έρευνα να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός των ντρόουν που μας ενδιαφέρουν και να αφιερωθούμε αποκλειστικά και μόνο στα μη επανδρομένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για επικίνδυνους στρατιωτικούς, τρομοκρατικούς και άλλους τους κακόβουλους σκοπούς. Άρα να στρέψουμε ε, το δυναμικό μας και τις δυνάμεις των ε, ε, δυνάμεων τάξης προς τα ντρόν που χαρακτηρίζουμε ως εχθρικά. Αυτή λοιπόν είναι η στρατηγική και η φιλοσοφία μας. Βασιστήκαμε σε δύο πυλώνες. Πρώτον το κανονιστικό ρυθμιστικό πυλώνο που ισχύει για την εθνική επικράτεια και όχι για τις επιχειρήσεις μας στο εξωτερικό. Και δεύτερος πυλώνας είναι η εξουδετέρωση των ε, drone εξουδετερήσει που ισχύει και στην εθνική μας επικράτεια αλλά και στις επιχειρήσεις μας στο εξωτερικό για το στρατιωτικό μας σκέλος. Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν από πλευράς κανονιστικής ισχύει η νομοθεσία, ισχύει η νόμος στη Γαλλία εδώ και δύο χρόνια που ε, καλεί τους πλοηγούς των μη επαδρομένων αεροσκαφών και, τον, και τους κατασκευαστές να ε, τηρήσουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρέπει να υπάρχει ε, ε, υποχρεωτική κατάρτιση και εκπαίδευση και για τους επαγγελματίες και για τους ερασιτέχνες. Πρέπει όποιος πετάει ντρό να καταχωριστεί σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα με τα στοιχεία του και να καταχωρήσει και το δικό του ντρόν το οποίο πρέπει να εκπέμπει ηλεκτρονικό σήμα αναγνώρισης και ταυτοποίησης για να ξέρουμε ποιο είναι αυτό το ντρόν που πετάει και αν ανήκει στον κατάλογο με τα συνεργαζόμενα ντρόν που έχουμε εμείς συντάξει, αν είναι ένα από τα δικά μας τα οποία αναγνωρίζουμε και τα θεωρούμε θεωρούμε ότι συνεργάζονται και πρέπει να έχει και φωτεινό, ε, φωτεινή λιχνία αναγνώρισης για να φαίνεται και τη νύχτα και να μην είναι αόρατο. Αυτά ε, εν ολίγης περιλαμβάνονται στην ομοθέσια Και βεβαίως συμβάλλουμε ε, στη σύνταξη και στην ομοπαρασκευαστική διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι γαλλικές αρχές τίνουν προς το ευρωπαϊκό μοντέλο για να έχουμε ομοιομορφία μόλις ψηφιστεί και υιοθετηθεί ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Συμβάλλουμε δηλαδή στη διατύπωση και στη σύνταξη αυτού. Ένα δεύτερο έργο που φέραμε σε πέρασα ε, ε, εκ παραλίλου είναι η ταυτοποίηση και η αναγνώριση του ντρόν που θεωρείται εχθρικό, που δεν συνεργάζεται και ο τρόπος με τον οποίο θα εξουδετερωθεί. Η γαλλική κυβέρνηση χρηματοδότησε σε ύψος 1,4 εκατομμύρια ευρώ τρία project, τρία έργα τα οποία παρουσιάστηκαν σε δημόσια συνεδρίαση ε, και τα οποία επελέγησαν από τα διάφορα υπουργεία για το στρατό, για τις ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις αγόρασαν ένα από αυτά τα συστήματα και το αναπτύσσουν αυτή τη στιγμή εντός ε, τους. Μπορούν να αναγνωρίσουν, να ανοιχνεύσουν τα ντρόν αυτόνομα, μπορούν να τα ταυτοποιήσουν, γιατί είναι δύσκολο να ταυτοποιήσει κανείς να αναγνωρίσει ένα ντρόν και να πει ότι δεν είναι όχημα ή δεν είναι πουλί, γιατί έχει περίπου το ίδιο σχήμα, και μετά πώς το εξουδετερώνει. Χωρίς να προδώσουμε λοιπόν στρατιωτικά μυστικά, η εξυδετέρωση των drone γίνεται μέσα από αυτό το οποίο ονομάζουμε στα γαλλικά brouqueur, δηλαδή μηχανήματα τα οποία παρεμβάλλονται και ε, το μπερδεύουν και το οδηγούν αλλού. Τώρα, σε εθνικό επίπεδο, οι εργασίες ε, συνδέονται άμεσα, δηλαδή οι εργασίες στο κομμάτι το πολιτικό της κοινωνίας και στο κομμάτι το στρατιωτικό. Με τον ίδιο τρόπο εφαρμόζονται δηλαδή όλες οι διαδικασίες και από τη Γαλλική Αστυνομία και από τη Γαλλική Χωροφυλακή, έτσι όπως εφαρμόζονται και από τις Γαλλικές Ενοπλές Δυνάμεις, στη δική μας εθνική επικράτεια. Επομένως, συνεχίζονται οι εργασίες μας, συμπερασματικά να πω, ε, ως προς το κανονιστικό σκέλος, ως προς την νομοθεσία και τη ρύθμιση και συμβάλλουμε και στην Ευρωπαϊκή Νομοπαρασκευαστική Διαδικασία. Το δικό μας εθνικό πλαίσιο, το νομικό, το έχουμε διαμορφώσει, δεν μένουν πολλά να γίνουν. Συμβάλλουμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Νομοθετική Διαδικασία Χρηματοδοτούμε επίσης έργα έτσι ώστε οι κατασκευαστές να συλλάβουν μέσα καταπολέμησης των ντρόν, τα οποία θα είναι διαφορετικά από αυτό το μπουγιάζ, από αυτό το μπέρδεμα, το οποίο είναι λειτουργικό, είναι αποτελεσματικό, ε, το, το μέσο των παρεμβολών δηλαδή. Έχουμε μηχανήματα που παρεμβάλλονται και κάνουν παρεμβολέ στα ντρόν και τα οδηγούν αλλού και δεν τα αφήνουν να πετύχουν το στόχο του. Υπάρχουν όμως όρια σε, αυτό το, σε αυτή την τεχνική δυνατότητα των παρεμβολών. γιατί υπάρχουν και μία παδρομένα αεροσκάφη που έχουν αυτόνομη δυνατότητα πλοήγησης και δεν χρειάζεται να παίρνουν την πορεία τους από δορυφόρο ή από εξωτερικό πομπό και ξέρουν μόνα τους που να πάνε και άρα δεν μπορούμε να, τα, να κάνουμε παρεμβολές και να τα μπερδέψουμε. Επομένως χρηματοδοτούμε την έρευνα για νέες τεχνικές καταπολέμησης των μη επανδρομένων αεροσκαφών και ελπίζουμε να ακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και να μην μείνουμε πίσω. Αυτά προς το παρόν κυρία Πρόεδρε, παραμένω στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Κρατήσατε και το χρόνο που είχε προβληθεί για σας. Ε, θα συνεχίσουμε και μετά, στο τέλος, ε, θα κάνουμε τη συζήτηση αφού ακούσουμε και τις τρεις εισηγήσεις. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ρόμπερτ Μορέι, ο οποίος ε, ασχολείται με θέματα παρακολούθησης, αναγνώρισης στον σχετικό τομέα στο ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σταθώ και σε κάποια από τα σημεία τα οποία ανέφερε και ο προηγούμενο ομιλητή και τα οποία θεωρώ ενδιαφέροντα. Ζητήματα ε, διαχείριση ενέργεια κυκλοφορία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα όταν έχουμε να κάνουμε με τα μη πανδρομένα αεροσκάφη. Είναι βέβαια αρκετή η ορολογία. Ε, εγώ θα αναφέρω μόνο τα drones για να συνοηθούμε. Και εγώ θα το εξετάσω από πλευρά τη καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Και φυσικά από στρατιωτική σκοπιά. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε τα βασικά οικονομικά ωφέλη των μικρών αυτών αεροσκαφών για την Ήπειρό μας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Ήδη το βλέπουμε όταν μιλούμε για την ε, αλυσίδα εφοδιασμού και την ευρεία διάδοση ε, των μικρών αυτών αεροσκαφών ε, στους εθέρες μας, καθώς αναπτύσσονται και άλλες τεχνολογίες, όπως το 5G, η αυτοματοποίηση, οι αλγόριθμοι στην ε, τεχνητή νοημοσύνη. Επομένω, πρέπει να είμαστε αρκετά ευέλικτοι και ανοιχτόμυαλοι ε, σε ό,τι αφορά τις, την αντιμετώπιση των απειλών και της κατάχρηση αυτών των τεχνολογιών. Το όνομα μου είναι Robert Murray. Εγώ εργάζομαι λοιπόν στο επιτελείο του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ και θα σας παρουσιάσω ορισμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη από στρατιωτική ε, σκοπιά και από πλευρά τη συμμαχία μα, ιδίω ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη δημοκρατία. Και εν συντομία, θα θίξω και τι κάνουμε εμεί για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο στο ΝΑΤΟ. Να σα πω ευθύ εξ αρχή ότι ενώ τα drones ίσως ε, μετατοπίζουν ε, την προσέγγιση μας ό,τι αφορά το χαρακτήρα των συγκρούσεων και η σημερινή συνεδρίαση βασικά σε αυτές τις μετατοπίσεις εστιάζει, κατά τη γνώμη μου τα drones δεν μετατοπίζουν πραγματικά το χαρακτήρα ε, των συγκρούσεων και έτσι θεωρούμε ότι αυτές οι προσαρμογές είναι, αποτελούν μια ε, εξελικτική διαδικασία και όχι μια ριζοσπαστική μεταμόρφωση ε, των πολεμικών συγκρούσεων. Όπως ξέρετε, τα drones έχουν πολλές ε, μορφές και πολλά μεγέθη. Εγώ θα επικεντρωθώ στα μικρότερα αεροσκάφη που μας παρουσίασε και ο Κριστόφ προηγουμένω στις διαφάνειες. Αυτά μπορείτε να βρείτε και στο Amazon ή αλλού, σε, στο τόπους. Μπορούμε βεβαίως να συζητήσουμε και τα μεγαλύτερα αεροσκάφη, αν μου θέσετε τέτοιες ερωτήσεις στη συνέχεια. Βλέπουμε όμως ότι συχνά ε, είναι ε, θολά τα όρια μεταξύ των υβριδικών ε, συγκρούσεων, τρομοκρατικών απειλών και συμβατικών. Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς ποιοι είναι οι δράστες όταν έχουμε αυτές τις τεχνολογίες. Ο Κριστόφ ανέφερε πώς έχει η απειλή αυτή τη στιγμή, πολύ ωραία, δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ εγώ. Βλέπουμε όμως ότι έχουμε ένα συνδυασμό συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο και πιο συγκεκριμένα στη Συρία και στο Ιράκ ιδιαίτερος. Ε, υπάρχει συνδυασμός με ε, δραστηριότητες και ενέργειες προηγμένης τεχνολογίας. Οι τρομοκράτες, όλο ένα και περισσότερο, κάνουν κατάχρηση ε, και κακόβουλη χρήση των τεχνολογιών που υπάρχουν ε, για την προετοιμασία, το σχεδιασμό, την προετοιμασία και εκτέλεση ε, αυτών των επιθέσεων. Και οι επιθέσεις εγείρουν ερωτήματα για την ανθεκτικότητα και ετοιμότητα των εταίρων μας, στις πατρίδες μας δηλαδή, έναντι αυτών των κοινών απειλών και οδηγεί σε ενέργειες όπω αυτέ που ανέφερε ο Κριστόφ από γαλλική άποψη, την ανάπτυξη στρατηγικών και ούτω καθεξή. Αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ε, στο σύνολο των χωρών του ΝΑΤΟ. Όμως βλέπουμε ότι οι τρομοκράτες ε, εκμεταλλεύονται και προσαρμόζουν αυτή την εμπορική χρήση τεχνολογία. Και είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι η στρατική ικανότητα. Και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τον ΝΑΤΟ και τους συμμάχους ε, να διασφαλίσουν την ε, διαθεσιμότητα κατάλληλων αντιμέτρων εγκαίρως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φυσικά αντίμετρα. Τα ανέφερε και κάποια από αυτά, μάλλον ο Κριστόφ προηγουμένω. Και γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλειά σε όλη τη συμμαχία. Όμω μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε βρει ακόμα τη χρυσή τομή για την πρόληψη, ε, την αποτροπή τέτοιων επιθέσεων και την αποκατάσταση τυχών ζημιάς απαιτείται μια πολυεπίπεδη αντιμετώπιση ε, με συγκέντρωση προσπαθειών από όλους τους συμμάχους, ε, τη βιομηχανία, την, τον ακαδημαϊκό χώρο και ούτω καθεξής. Εξαιτία τη πιθανής εξέλιξης αυτής της απειλής από την κακόβουλη χρήση των εναέριων ε, αεροσκαφών drones σε μια πιο γενικευμένη ε, χρήση ε, νέων τεχνολογιών που θα περάσουμε πλέον και στις ε, χερσαίες, και σε χερσαία τέτοια ή θαλάσσια σκάφη είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως από στρατιωτικής άποψη. Ανέφερα λοιπόν ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και οι εθνικές υπηρεσίες ε, καταβάλουν πολύ σημαντικέ προσπάθειε για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών. όμω το ΝΑΤΟ ω οργανισμό αυτή τη στιγμή δεν έχει ένα ε, συνολικό σφαιρικό πλαίσιο που να συντονίζει αυτέ τι προσπάθειες για την αντιμετώπιση ιδίω αυτών των μικρών drones. Όμω είμαστε πολύ κοντά στην οριστικοποίηση ενός ε, σχεδίου, πλαίσιο ε, για την αμυντική μας προσπάθεια και θα το υιοθετήσουν και οι Υπουργοί ε, Αμήνης ε, στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Οι ικανότητες καταπολέμησης των drones όμως δεν ακολουθούν την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων που έχουμε παρατηρήσει στα drones, ιδίως ό,τι φορά τα μικρά εμπορικής χρήσης drones. Ε, βλέπουμε το πώς ε, λειτουργούν τα αντίμετρα σε διάφορα περιβάλλοντα και σε διάφορες ε, μορφές στρατιωτικών επιχειρήσεων ή το πώς η απόδοσή τους για συγκεκριμένες απειλές μπορούν να ληφθούν υπόψη για άλλη χρήση. Οποιαδήποτε σωστή αντιμετώπιση των drones από στρατιωτική άποψης θα είναι μια προσέγγιση συστήματος συστημάτων. Δεν έχουμε βρει λοιπόν ε, τη μαγική λύση ακόμα. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε τη διαλειτουργικότητα και να μην ε, αποτρέπουμε, να μην ε, παρεμποδίζουμε τις φιλικές ενέργειες. Γι' αυτό και το σχέδιο δράσης μας επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς τομείς. Δημιουργία ενός οικοσυστήματος μεταξύ συμμάχων ε, με αξιοποίηση εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας από άλλες κοινότητες όπως η αντιμετώπιση των εκλεκτικών ε, ε, μηχανισμών. Δεύτερον, πλήρης αναθεώρηση πολιτικής, επανεξέταση της σημερινής, εντοπισμός κενών και κάλυψή τους με νέες τακτικές, νέες διαδικασίες ε, που θα πρέπει να έχουν οι δυνάμεις μας ε, επιτόπου. Η ανάπτυξη προτύπων. Όλα θα πρέπει να λειτουργούν ε, απρόσκοπτα, το οποίο είναι εύκολο να το λέμε, δύσκολο να το κάνουμε πράξη. Και να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με ταχύς ρυθμούς. Θέλουμε να επιταχύνουμε το ρυθμό της αντιμετώπισης μας. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να επισημάνω ότι στρέφουμε το βλέμμα προς το μέλλον. Αρχίσουμε να βλέπουμε τεχνολογίες ε, όπως ε, το 5G, ε, τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον είναι ευρείας χρήσης, εκτύπωση 3D και διάφορες άλλες τεχνολογίες. Επομένω και οι τεχνολογίες στα drones μόνο να αυξηθεί πρόκειται και μάλιστα με ε, ταχύς ρυθμούς. Παρότι αυτό αποτελεί πρόκληση από πλευράς ε, ασφάλειας και άμυνας, δεν πρέπει να ξεχνούμε και τα τεράστια οικονομικά ωφέλη αυτής της τεχνολογίας. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Αξιοποίηση των οικονομικών ωφελών, αλλά και από την άλλη ε, ασφάλεια και προστασία των ε, δυνάμεών μας και του πληθυσμού φυσικά είναι μια μεγάλη πρόκληση. Όμως, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κακόβουλη χρήση αυτή τη τεχνολογία. Γι' αυτό και στο ΝΑΤΟ επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας ακριβώς σε αυτό το σημείο, για, την, για να έχουμε αντίμετρα και τεχνολογία που να καταπολεμά αυτή την ε, τεχνολογία όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Πολύ ωραία. Δίνω το λόγο στον επόμενο εμπειρογνώμονά μας, ε, ο οποίος είναι από το Fisher Institute ε, για στρατηγικές μελέτες ε, στο Ισραήλ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την πρόσκληση και τη συζήτηση που γίνεται, η οποία βέβαια είναι πολύ μεγάλη σημασία. Μου ζητήθηκε να μιλήσω εβραϊκά και θα το πράξω. Λέγομαι Ταλιμπάρ, είμαι από το Ινστιτούτο Φίσερ του Ισραήλ ε, και συμφωνώ απόλυτα με τους ε, προαλήσαντες σχετικά με τις προκλήσεις που είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν στο μέλλον. Ε, θα ήθελα να εκφράσω κάποιες δικές μου σκέψεις, αυτών όσων ελέγχθησαν και θα ήθελα επίση να υπογραμμίσω ότι εδώ στην Ευρώπη βλέπουμε να υπάρχουν παραδείγματα των ε, μικρών ντρόουν ενός ε, που το χειρίστηκε ένας ε, δημοσιογράφος και σχεδόν προσγειώθηκε μπροστά στο βήμα που μιλούσε η κυρία Μέρκελ. Αυτό έγινε πριν από λίγο καιρό. Βέβαια ήταν καλόβουλη πράξη. Στο Ισραήλ υπάρχουν πάρα πολλές ε, περιπτώσεις επιθέσεων με drones από το 2006. Ορισμένες από αυτές ε, είχαν ε, εκτοξευτεί από το Λίβανο, από τη Χεσμολά και πολύ πρόσφατα είχαμε ένα μη επαντρωμένο υπτάμενο όχημα, ένα με τέσσερις έλικες ήταν αυτό, ένα quadcopter και ξεκίνησε από το Ιράν. Θεωρείται λοιπόν ότι είναι ένα επιθετικό ντρόν το οποίο διείσδησε στον ενάριο χώρο του Ισραήλ και καταρρίφθηκε από τον ε, Ισραηλινό στρατό. Η απειλή λοιπόν είναι πραγματική και έχουμε τα drones και με τι σταθερές πτέρυγες, αλλά και εκείνα με, τις, με τους όπως έχουν τα ελικόπτερα και τα δύο αποτελούν κίνδυνο και καθίστανται όλο και πιο επικίνδυνα και εξαπλώνονται μάλιστα. Βλέπουμε να χρησιμοποιούνται σε διάφορε συγκρούσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Χρησιμοποιούνται αυτά τα οχήματα τα οποία καθίστανται όλο και πιο εξελιγμένα. Πρέπει λοιπόν να διαφοροποιούμε ανάμεσα σε απειλέ, σε καιρό ειρήνης και σε καιρό πολέμου. Και πρέπει σε καιρό ειρήνης να συνεργαζόμαστε με τους κατασκευαστές των ε, ε, μη επανδρομένων ε, οχημάτων, να παρεμποδίζουμε την υπερπτήση τους από μη καθορισμένες περιοχές. Παραδείγματος χάρη στη, στο Ισραήλ είχαμε διείσδυση από ντρόν και από μη επανδρομένων υπτάμενων οχημάτων, των UAV. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε στο ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε και με το στρατό και να βρούμε και σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Αυτός είναι ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Τώρα, οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των μη επανδρομένων υπτάμενων οχημάτων, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στην κλασική αντιμετώπιση των αντιεροπορικών επιθέσεων με ε, στρατεύματα εδάφους. Ίσως θα μπορούσα να σας δείξω ορισμένες διαφάνειες που να σας ενδιαφέρουν, γιατί εξετάζουμε όχι μόνο το θέμα των ντρόν αλλά και το θέμα των ε, ε, πυρομαχικών και τη μετάβαση από πολύ πρόχειρο ε, πρόχειρο εξοπλισμό και πυρομαχικά στην περίπτωση αυτή που μεταφέρονται από το ISIS στη Συρία, στο Ισραήλ και εδώ βλέπουμε ε, χειροβομβίδες ε, εξελιγμένες τεσσάρων χιλιοστών. Βλέπουμε όμως και άλλες ε, βόμβες που είναι κατασκευασμένε, είναι με ένα είδο βλημάτων τα οποία κατασκευάζονται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Είναι αυτός πολύ εξοπλισμένο ε, εξοπλισμό και πυρομαχικά. Αυτό βέβαια ε, είναι ένα επίσης ε, πολύ πρόχειρο όπλο το οποίο κατασκευάζεται στο Ιράκ αλλά και στη Συρία. Και αυτά κατασχέθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ. Εδώ βλέπετε μία εικόνα η οποία δημοσιεύτηκε από τον ISIS. Ε, βλέπετε τη βόμβα, από κάτω βλέπετε το τάγκ και ε, διάφορα άλλα στρατιωτικά οχήματα, τα οποία ένα εξ αυτών καταστράφηκε από μία μικρή βόμβα, την οποία εκτόξευσε, υποτίθεται, ένα ντρόν παιχνίδι. Ο συνάδελφός μου από τη Γαλλία είπε ότι Είδαμε και την επίθεση στην αεροπορική βάση Χεμιμίμ στη Συρία, όπου χρησιμοποιήθηκαν τα μη παντρωμένα αυτά οχήματα για να αντιμετωπιστούν, να να υπάρξει επίθεση στις ρωσικές δυνάμεις. Ε, βλέπουμε ε, το 3D, ε, την κατάτμιση αλλά οφείλω να επισημάνω ότι η ζημιά δεν ήταν τόσο μεγάλη. Αυτό είναι ένα αεροσκάφο το οποίο δέχτηκε την επίθεση από αυτές τις μικρές βόμβες. Αυτά για σήμερα. Αύριο όμω, αυτά μπορεί να συμβούν σε ένα μη στρατιωτικό αεροδρόμιο και μπορείτε να κατανοήσετε τι θα συμβεί αν υπάρξει μια τέτοια επίθεση σε ένα πολυσύχναστο αεροδρόμιο με ε, πολλούς επιβάτες σε μη στρατιωτικά αεροσκάφη. Η τάση λοιπόν είναι να γίνονται τα όπλα όλο και πιο αποτελεσματικά. Εδώ βλέπετε την κεφαλή από ε, ένα πύραυλο που και αυτός ε, έπεσε στη Συρία. Εντοπίστηκε στη Συρία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα ε, κατευθυνόμενο πύραυλο για να πλήττονται θωρακισμένα και θα ήθελα να σας δείξω κάποιες τάσεις που επικρατούν στην κατασκευή Αυτά τα χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά οι τρομοκράτες ε, και τώρα πλέον ε, γίνεται μια τεχνολογία η οποία εξαπλώνεται όλο και περισσότερο. Άλλο θέατρο επιχειρήσεων είναι βέβαια η εμένη. Βλέπουμε ότι εκεί υπάρχουν πολύ μικρά ε, μη επανδρομένα αεροσκάφη στις επιδρομές των Χούτι και παρεπιπτόντος αυτό εισήχθη Δηλαδή, στόχος ήταν να πληγούν κάποιοι στόχοι στην Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και παρεπιπτόντος, αυτό είναι ένα drone το οποίο προήλθε από το Ιράν. Και το έχουμε δει και στο Ισραήλ. Δεν θα ήθελα να ε, μιλήσω διαμακρών στο θέμα της εξαγωγής ε, των ντρόν και των μη πανδρομένων οχημάτων από το Ιράν, αλλά βλέπετε εδώ αυτή την διαφάνεια όπου το Ιράν χρησιμοποιεί ντρόν τα οποία ε, έχουν προέλθει από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα τα αντιγράφουν και τα πουλάνε σε άλλες χώρες. Εάν λοιπόν μιλάμε για προϊόντα που μπορεί κανείς να αγοράσει ε, στο διαδίκτυο ή οπουδήποτε αλλού αυτό σημαίνει ότι μερικές φορές ε, τα μη παντρωμένα οχήματα θα μπορούσαν να πέσουν στα χέρια οποιοδήποτε και να αποτελέσουν απειλή για το μέλλον. Ως εκ τούτου πρέπει να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα και αυτό είναι το τελευταίο γεγονός όπου χρησιμοποιήθηκαν τα μη παντρωμένα υπτάμενα οχήματα, τα UAV ε, στο Ισραήλ κατερρίφθη, είχε εκτοξευτεί από τη Συρία. Και πρόσφατα εκτοξεύτηκε από οι Ιρανικές δυνάμεις ε, κατά στόχων Κούρδων στο Ιράκ. Η απειλή λοιπόν είναι πραγματική. Αυτά είναι τα συμπεράσματά μας. Και δεν έχουμε ακόμα όλες τις απαντήσεις. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο και τα UAVs ε και τα drones και θα μπορούσε όλο αυτό να προσφέρει στον επιτιθέμενο την ασπίδα της ε, ανωνυμίας, γιατί όλα αυτά μπορεί κανείς να τα χειριστεί ε, μέσω δορυφόρου με απόλυτη ανωνυμία. Η δική μου άποψη επί του θέματος είναι ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε καταρχήν το πρόβλημα, να προβλέψουμε και να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Η άμβλυνση του ε, προβλήματος θα μπορούσε να γίνει με κυβερνοεπιθέσεις, ε, με επιθέσεις ε, hard kill, αντιαρματικές, με πυράβλους όπως το έχουμε κάνει ήδη αρκετές φορές και όσον αφορά τώρα τις προκλήσεις SWORM, αυτό κατά την άποψή μου πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα Πολλές φορές ε, βλέπουμε αυτή τη θαυμάσια εικόνα των ντρόουν ε, στον ουρανό με πολύ ωραία φώτα τη νύχτα, αλλά το να γίνονται αυτά τα σμήνη των ντρόουν πάνω σε πυρηνικούς σταθμούς ή πάνω σε στρατιωτικές βάσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να το περιορίσουμε και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Και όσον αφορά τώρα το τελικό μου συμπέρασμα είναι πριν από δύο εβδομάδες στην Κίνα είχαμε μια μεγάλη έκθεση αεροσκαφών του τομέα όπου κινέζικες εταιρείε παρουσίασαν τη νέα εξέλιξη των ντρόν που είναι ε, ε, εξοπλισμένα με πολύ προχωρημένους και εξελιγμένους αντιαρματικούς πυράβλους, με εκτοξευτήρες, με όλο αυτόν τον εξοπλισμό. Είδαμε λοιπόν αυτά τα ντρόουν για πρώτη φορά να χρησιμοποιούνται στο χώρο της τρομοκρατίας, αλλά τώρα είναι κάτι που μπορεί κανείς και να αγοράσει. Όλα αυτά σημαίνουν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο αυτά τα οχήματα στο μέλλον. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το θαυμάσιο άγαλμα που λέει εδώ είσαστε έτοιμος για την πρόκληση. Ναι, αλλά όχι επαρκώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ε, τελική εικόνα που νομίζω ότι ε, είναι και μια πάρα πολύ καλή κατακλίδα όλων αυτών που ελέγχθησαν. Γιατί έχουμε μια τεράστια βεντάλια των προκλήσεων ε, τόσο τεχνικής όσο και νομικής και ηθικής μορφής. Εγώ έχω συγκρατήσει τη λέξη απειλή. Είναι η λέξη που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από όλες τις άλλες. Και παρότι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ανώτερα στελέχη και προβεβλημένους ε, εμπειρογνώμονες, έχω την εντύπωση ότι οι απειλές που αναφέρθηκαν, που παρουσιάστηκαν και οι απαντήσεις που εδότησαν δεν είναι ικανοποιητικέ, δεν ταυτίζονται. Γιατί εξακολουθώ να έχω κατά αυτό που είπατε, ότι η απειλή προχωράει και εξελίσσεται πολύ περισσότερο από τις δυνατότητες που υπάρχουν για να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εσά στους συναδέλφους μου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ο κύριος Γκάλερ έχει ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που είπατε, πολύ ενδιαφέροντα. Καθαρά έτσι αυθόρμητα, όταν μιλάγατε κύριε Ιμπάρ, σκέφτηκα το εξή. Ε, είχα την εντύπωση ότι κάτι δεν πρέπει να έκαναν καλά το Ισραήλ και οι ΗΠΑ. Κάτι έκαναν στραβά. Το να είναι τώρα το Ιράν σε θέση να κατασκευάζει μιμούμενο αυτό το drone, ε, κάτι δεν πήγε καλά. Μα τι κάνατε, δεν ε, εντάξατε έναν μηχανισμό αυτοκαταστροφής ή οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε στο τέλος να μπορείτε να παρακολουθείτε το τι ακριβώς κάνουν οι Ιρανοί με όλα αυτά. Ίσως βέβαια να στείλατε ένα δόλωμα, να το κάνατε επίτηδες, να το στείλετε στους Ιρανούς, ακριβώς για να το μιμηθούν και να το κατασκευάσουν. Μπορεί να υπάρχει και αυτή η άποψη εθίγησαν πάρα πολλά θέματα. Εγώ ένα θέμα θέλω να επισημάνω. Πρόκειται για την κοινή χρήση του ε, εναέριου χώρου, ο οποίος χρησιμοποιείται και για στρατιωτικούς και για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Αυτό που ενδιαφέρει τώρα είναι στον δικό μας, τον ευρωπαϊκό χώρο, να επιτυγχάνουμε το συντονισμό. Και για να το πετύχουμε αυτό Θεωρώ ότι είναι σωστό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, ο οργανισμός αυτός ε, να συμπεριλαμβάνει στην όλη συζήτηση και τις ε, στρατιωτικές ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνομαι στους εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με πρακτικά θέματα για να μας πούν τελικά τι γίνεται. Ε, όταν έχουμε καιρό ειρήνης, όταν δεν πρόκειται για στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά όταν πρόκειται για την κανονική απλή χρήση από πλευράς ε, ενόπλων δυνάμεων. Υπάρχει εναρμονισμός και συντονισμός των δομών με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι δυνατόν από ένα και μόνο σημείο να υπάρχει η απόλυτη καθοδήγηση. Στα νέα προγράμματα της ε, ΠΕΣΚΟ, της ε, ε, μόνιμης αυτής δομής συνεργασίας. Έχουμε ορίσει το ότι στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, στο Single European Sky, θα πρέπει να υπάρχει διαρθρωμένη συνεργασία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω, στο βαθμό που μπορείτε και εσείς να απαντήσετε, τι πιστεύετε επ' αυτού. Κατά τα άλλα, Θέλω να κάνω άλλη μία ερώτηση που αφορά στις κυβερνοαπειλές. Παραδείγματο χάρη, η αποστολή δεδομένων και η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα σε δεδομένα και ντρόν. Μπορούμε αυτά να τα προστατεύσουμε έναντι των ε, επίδοξων ε, εχθρών. Υπάρχει κάποιος μηχανισμός άμυνα σε σχέση με τα δεδομένα που επικοινωνούν με τα ντρόν είμαστε σε επίπεδο να αντιμετωπίσουμε τις απειλές. Και επίση, ποια είναι ακριβώς η συνεργασία που να αφορά πέρα από το ΝΑΤΟ και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνεργασία και με το Ισραήλ. Η συνεργασία με το Ισραήλ είναι σε οικονομικό και βιομηχανικό επίπεδο ή μήπως η συνεργασία αφορά και την ανταλλαγή πληροφοριών για λόγους ε, πολιτικής και ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν επιθυμεί κάποιος άλλος ε, να λάβει το λόγο, να υποβάλει ερωτήματα. Αυτή η τεχνική διάσταση του θέματος, ε, από ό,τι φαίνεται σας φόβησε, αυτή την εντύπωση έχω, είναι εκφοβιστική. Και εγώ, πέρα από την ιδιότητά μου της Προέδρου, έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις και έχω να κάνω και κάποια σχόλια. Θα πω λοιπόν το εξής. Εγώ είμαι συγγήτρια και για θέματα ελέγχου ε, εξοπλισμών και εξαγωγών όπλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που με απασχολεί λοιπόν είναι πώς μπορούμε να έχουμε έναν αποτελεσματικό έλεγχο εξαγωγής όπλων. Ο έλεγχος εξαγωγής όπλων αφορά ε, προφανώς ε, και το θέμα των τεχνικών δυνατοτήτων. Όχι μόνο τα όπλα. Ίσως λοιπόν έχετε κάτι να μας πείτε από αυτού. Παραδείγματο χάρη, αυτό το θέμα της μεταφοράς δυνατοτήτων και αυτό της κατασκευής των ντρών από το Ιράν. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν ερωτήματα στον τομέα. Κατόπιν έγινε λόγος για οικονομική χρήση. Τώρα μιλάμε για επανδρομένα, μάλλον εξοπλισμένα συστήματα drone με όπλα και αυτό που με ενδιαφέρει είναι κατά πόσον αυτά τα εξοπλισμένα ε, με όπλα drone, κατά πόσον ε, αυτά τα νέα drone ε, δημιουργούν ένα πρόβλημα και από πλευράς οικονομικής. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει κατ' ουσίαν πρόβλημα και όσον αφορά τον ε, εντοπισμό των ε, χρηστών. Ε, πρόβλημα υπάρχει και στο πού ακριβώς ορίζονται τα όρια. Πώς μπορεί κανείς να παρέμβει και αν μπορεί να παρέμβει εφόσον εντοπίζεται ένας κακόβουλος χρήστης. Παρόλα αυτά όμως ε, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια όρια των δυνατοτήτων παρέμβασης. Έχοντας κατά νου το γεγονός ότι μια ζημιά η οποία έχει προκληθεί, κατ' ουσίαν αυτή η ζημιά μπορεί να σημαίνει απώλεια πολλών ανθρώπινων ζώων και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε πολλές ακροάσεις ε, ε, και σχετικά με το θέμα το πώς μπορούν οι άνθρωποι να συνεχίσουν την κανονική τους κοινωνική ζωή. Ε, έχουμε λοιπόν ένα ψήφισμα ε, που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία και απορρίπτει τα αυτόνομα οπλικά συστήματα και την ε, δολοφονία με αυτά τα συστήματα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω και εγώ να θέσω το εξής ερώτημα. Αυτά τα συστήματα τα οποία έχουν θανατηφόρες δυνατότητες ίσως θα πρέπει να απογορευτούν αυτά τα συστήματα και αυτοί οι εξοπλισμοί. Γιατί θα πρέπει να έχουμε κατά νου περιπτώσεις όπου τα συστήματα αυτά ούτε να εντοπιστούν μπορούν, να αναγνωριστούν, αλλά ούτε και να αντιμετωπιστούν. Και θα πρέπει να σκεφτούμε το τι μπορεί κανείς να κάνει σε σχέση με αυτά τα συστήματα και τους εξοπλισμούς που υπάρχουν. Αυτά είχα να πω και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους εμπειρόγνωμονές μας, εκτός αν εσείς θέλετε να υποβάλλετε συμπληρωματικές ερωτήσεις. Από ό,τι βλέπω όχι, ως εκ τούτου δίνω το λόγο στους εμπειρογνώμονες με την ίδια σειρά που αρχίσατε και λάβατε το λόγο, γιατί κάποιος από εσά νομίζω είπε και ότι θέλει να φύγει νωρίτερα. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις ερωτήσεις σας. Δύσκολα θα μπορέσω να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις, γιατί νομίζω ότι και οι άλλοι συνάδελφοι είναι πολύ κατάλληλοι να απαντήσουν. Κυρίως ο συνάδελφος από το Ισραήλ θα θέλει σίγουρα να απαντήσει για το Ιράν. Με ρωτήσατε όμως για την αρχή του UTM και πώς το συλλάβαμε, πώς τη συλλάβαμε αυτή την ιδέα. Ξέρετε πιο πολλά για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Ωστόσο, έχουμε έργα και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να συμφιλιώσουμε τις ε, εναρείς κυκλοφορίες μη επανδρομένων αεροσκαφών με την ε, κυκλοφορία ε, των ε, κανονικών, επιβατικών, εμπορικών και άλλων αεροσκαφών για να υπάρχει καλύτερη κυκλοφορία, για να μην υπάρχουν συγκρούσεις και για να προάγουμε τις υπηρεσίες που προωθούν τα ντρόουν. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 στο Παρίσι υπάρχει ένα project για την προσέγγιση μεταξύ αεροδρομίων και ε, αθλητικών εγκαταστάσεων ε, με ε, drone να μεταφέρονται οι επιβάτες μεταξύ ε, με τη βοήθεια των drone και με τη βοήθεια των ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Στη Τσεχία υπάρχει το AirMap, ένα project για την πρώτη υπηρεσία UTM που έχει αναπτυχθεί ε, και στην Ελβετία και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχουν δηλαδή κάποια έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα του συντονισμού των κινήσεων. Όλα αυτά γίνονται με συνεργατικό τρόπο και μη, με μη συνεργατικό. Όλα αυτά ελπίζω ότι θα συνενωθούν και θα συγχωνευτούν βάσει του UTM στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό όταν ολοκληρωθεί και αυτό το έργο. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σωστά υπογραμμίσατε τη δυσκολία εντοπισμού και αναγνώρισης και ταυτοποίησης των χριστών. Και αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της γαλλικής νομοθεσίας και της ε, ε, νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούμε από το χρήστη να καταχωρήσει την ταυτότητά του. Παρόλο που μπορεί να βάλει ψεύτικα στοιχεία, αυτά τα στοιχεία τα συγκρίνουμε με τα εθνικά αρχεία που τηρούν οι αστυνομικές αρχές για να αναγνωρίσουμε ε, κάποιον τον οποίο ε, ο οποίος είναι ήδη γνωστός στις αστυνομικές αρχές της χώρας, με την κακή έννοια του όρου βεβαίως. Και αυτό είναι στον πυρήνα της ε, ε, του κανονισμού, του νομοθετικού κειμένου. Ένα άλλο ερώτημα ήταν το εξή. Μήπω δεν πρέπει να απαγορευτεί, μήπω πρέπει τελικά να απαγορευτεί η χρήση των μη επανδρομένων αεροσκαφών για εμπορικού σκοπού, γιατί μπορεί να υπάρξει παρέκκληση από τη χρήση τους και να προκληθούν πολύ σοβαρά γεγονότα και που θα επιφέρουν και το θάνατο πολλών ατόμων. Εγώ πιστεύω πω όχι. δεν μπορούμε να τα απαγορεύσουμε. Γιατί παραμένει ένα παιχνίδι, μια ψυχαγωγική δραστηριότητα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κακόβουλο σκοπό, παραμένει όμως ένα παιχνίδι, άρα πρέπει να αναπτυχθεί ο οικονομικός κλάδος, δίνει νέες οικονομικές δυνατότητες, μιλούμε για την ατομική ελευθερία, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και μπορεί να υπάρξουν και χρήσεις πολύ σημαντικές και πολύ θετικές, τις οποίες ακόμα δεν έχουμε διανοηθεί. Το 2016 στην Νίκαια έγινε μια τρομακτική τρομοκρατική επίθεση. Κάποιος είχε νοικιάσει ένα φορτηγάκι και το έστρεψε εναντίον του πληθυσμού. Είχαμε πάρα πολλά θύματα. Καθημερινά νοικιάζονται φορτηγά στην Ευρώπη. Έγινε τεράστια δουλειά για να αναγνωριστεί ο δράστης των έχουμε κάνει τεράστια δουλειά δηλαδή για τις ενοικιάσεις οχημάτων προκειμένου να αποφύγουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις χωρίς να περιορίσουμε το δικαίωμα αυτό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ στον επόμενο μιλητή. Μάλιστα, ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα ερωτήματα και θα επανέλθω στην αρχή. Σε ό,τι αφορά τους ενιαίους ευρωπαϊκούς εθέρες, υπάρχει πολύ, πολύ μεγάλο συντονισμό μεταξύ του ΝΑΤΟ, του Eurocontrol και των υπολείπων ενδιαφερμένων μερών. Ιδίω ό,τι αφορά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Υπάρχει λοιπόν αυτό ο συντονισμό ε, αναμφίβολα. Ποια είναι η πρόκληση τώρα με τα μικρότερα ιδίω ε, drones που επεσήμανε και ο Κριστόφ είναι δυνατότητα για τα ραντάρ και τις τεχνολογίες μας να τα ανοιχνεύσουν, να τα εντοπίσουν. Γιατί φανταστείτε σε ένα τέτοιο αστικό περιβάλλον όπως είμαστε εδώ, ότι είναι πολύ κοντά μας, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο. Ε, για άλλα προγράμματα που έχουμε πολύ μεγαλύτερο υψόμετρο, τότε φυσικά και το Single Euro Sky και τα εθνικά συστήματα είναι πολύ σημαντικά. Αλλά όταν είναι χαμηλό το υψόμετρο σε ε, περιοχές ε, με μεγάλη συμφόρηση, αστικό περιβάλλον για παράδειγμα, τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό τους, πόσο μάλλον για την ταυτοποίησή τους. Στρατιωτική, drones έχουν κρυπτογράφηση τέτοιων δεδομένων. Αν είναι τώρα ε, ευάλωτοι στις κυβερνοεπιθέσεις, είναι όπως και οτιδήποτε άλλο. Όμως το επίπεδο ασφαλείας και κρυπτογράφησης είναι αρκετά υψηλό. Υπάρχει λοιπόν η καλύτερη δυνατή προστασία. Το ερώτημα τώρα για τη συνεργασία με το Ισραήλ το ΝΑΤΟ έκανε τον περασμένο μήνα ένα εργαστήριο ακριβώ για αυτό το θέμα. Την πρώτη μέρα λοιπόν συμμετείχε και το Ισραήλ μαζί με άλλους φορείς. Υπήρχε ε, ανταλλαγή πληροφοριών ε, όπως ήταν αναμενόμενο. Τώρα στρέφουμε προς τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων και τη τεχνική μεταφορά. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση, γιατί στον 20ο αιώνα, αν δείτε, πολλέ από τι τεχνολογικέ εξελίξει που πλέον θεωρούμε δεδομένε, όπω το διαδίκτυο, το GPS, ε, ε, η αύξηση τη υπολογιστική ισχύω, ε, προέκυψαν ουσιαστικά από τον στρατιωτικό και κυβερνητικό κλάδο. Στον 21ο αιώνα τώρα λοιπόν, με την κινητή τηλεφωνία, ε, τα drones, ε, την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά καλύπτονται από τον ε, τεχνολογικό κλάδο. Πώς θα τα ελέγξουμε όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο πλέον. Γιατί πλέον αυτή η τεχνολογία δεν προκύπτει από τον δημόσιο κλάδο, την κυβέρνηση, προκύπτει από τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει λοιπόν να το αναγνωρίσουμε αυτό. Και έτσι να δούμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρχει αυτή η τεχνολογική μεταβίβαση. Μίλησα για την ταυτοποίηση των drones, ότι είναι πολύ, κάτι το πολύ δύσκολο και σωστά είπε η Πρόεδρος ότι αυτό είναι πρόβλημα, σίγουρα. Δεν θα ήθελα να προτείνω ότι ως ε, σωστή λύση την απόλυτη απαγόρευση πρέπει να γίνει μια συζήτηση για τα πιθανά μακροοικονομικά ωφέλη όπως έγινε και με το διαδίκτυο και την υπολογιστική ισχύ και ούτω καθεξής. Και εκεί είναι πολύ σημαντικό το οικονομικό όφελος, υπάρχει όμως και σκοτεινή πλευρά. Αυτά πρέπει να διαχειριστούμε. Όμως νομίζω ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε ιδίως από στρατηγική σκοπιά, είναι να έχουμε ε, ένα χρονοδιάγραμμα ε, ανάπτυξης και εξέλιξης. Δηλαδή το χρονικό διάστημα που χρειαζόμαστε για να αγοράσουμε τον εξοπλισμό που θα αντιμετωπίσει αυτά τα drones είναι σε πολλές χώρες ε, μια δύσκολη διαδικασία. Και αυτό από μόνο την γιατί ακριβώς κινείται με τόσο ταχύς ρυθμούς η τεχνολογική εξέλιξη. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να μιλήσω εβραϊκά. Ε, Πρώτα απ' όλα, ένα ερώτημα το οποίο έθιξε η Πρόεδρος. Το ζήτημα του κανονιστικού πλαισίου. Πράγματι, μπορούμε να μιλήσουμε για περισσότερους με ένα ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε και τα έχουμε καταφέρει, αλλά αυτό δεν παρεμποδίζει ε, το παράνομο εμπόριο και διακίνηση αυτών των μηχανισμών. Πρέπει να κατανοήσετε ότι τα drones καταρχήν θεωρούνται παιχνίδια. Η τεχνολογία έχει έρθει και δεν πρόκειται να φύγει, θα εξελιχθεί περαιτέρω. Η τεχνολογία από μόνη της ε, δεν είναι καλή ή κακή όπως ένα μαχαίρι. Ε, στα χέρια ενός τρομοκράτη και στα χέρια ενός χειρουργού δεν έχουν την ίδια χρήση, ούτε το ίδιο αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι όσοι κινούνται πέραν του νόμου, πάντα θα βρίσκουν ε, τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία μας εναντίον μας. Και αυτό ισχύει με, σε οποιοδήποτε κλάδο για τις ε, κυβερνοεπιθέσεις. Πέραν τη συνεργασία που υπάρχει ήδη μεταξύ Ισραήλ και άλλων χωρών, ε, φαντάζομαι κατανοείτε όλοι ότι είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο και όλοι προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ε, ασφάλεια και προστασία όλων. Είτε μιλούμε για την έρευνα είτε ευρύτερα έχουμε να κάνουμε και με την ε, χρήση μη επανδρομένων αεροσκοφών ως πλατφόρμας που ε, μεταφέρει μηχανισμό υποκλοπών. Φανταστείτε τώρα, αν υπάρχει, ε, να υπάρχουν μερικά τέτοια drones πάνω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δημιουργούν ένα πλαστό δίκτυο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί πρέπει να δούμε ε, αν φτάνει μόνο η ε, νομική και νομοθετική αντιμετώπιση είτε ή αν πρέπει να στραφούμε προς τον κλάδο της τεχνολογίας για να βρούμε λύσεις. Υπόθηκε προηγουμένως ότι πρέπει να υπάρχει μία συμβίωση ε, αυτών των αεροσκαφών, των επανδρομένων και μη επανδρομένων. Είναι πρόβλημα αυτό στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ακόμα κανονιστικό πλαίσιο. Δεν μπορώ να πω ότι έχει λυθεί αυτό το ζήτημα. Ε, στο Ισραηλό Κοινοβούλιο υπάρχουν πολλές συνεδριάσεις ακριβώς για αυτό το, για το ζήτημα. δημοσιεύθηκε και μία ε, ιδιαίτερα εμπιστατωμένη έκθεση από την ελεγκτική αρχή για να εξετάσουμε ακριβώς ε, τις απειλές ε, των drones για την ενέργεια κυκλοφορία, τη δυνατότητα που έχουν αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη να ρίχνουν είτε δεσμίδες χρημάτων είτε παράνομων εμπορευμάτων. Αυτά δεν τα έχουμε λύσει ακόμα, ούτε εμεί ούτε γενικά στον κόσμο, για να έχουμε ασφαλείς εθέρες τελικά. Εν κατακλείδη, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε για την απειλή μη επανδρομένων ε, οχημάτων και εδάφους ε, και θαλάσσεις. Είναι κάτι το οποίο θα αρχίσει να μας απασχολεί όλο και περισσότερο από τρομοκρατικές οργανώσεις, από μη κρατικού ε, φορείς ε, και άλλες οντότητες που μπορούν να δημιουργήσουν και να αξιοποιήσουν τις τεχνολογικές δυνατότητες προς όφελός τους. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Hatte jetzt einer äh, diese eine Frage beantworten können um, äh, Κάτι δεν κατάλαβα. Ίσως δεν απάντησε κανείς το εξής ερώτημα, νομίζω. Εκτός και αν απατώμε. Δηλαδή, οι σύνδεσμοι με τα δικά μας ντρόουν μπορούν να υποστούν παρεμβολές έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις όπου χάθηκαν ντρόουν γιατί χάσαμε τον έλεγχό τους, γιατί οι συνδέσεις ε, είχαν υποστεί παρεμβολή από τον εχθρό. Μπορείτε να αποφύγετε οι εχθροί σας ε, να επηρεάζουν ε, την διασύνδεση δεδομένων με τα drone. Πώς ακριβώς ε, έχει το θέμα. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, δεν υπάρχει καταληκτική απάντηση, άσπρο-μαύρο, διαδική απάντηση θα έλεγα. Τα στρατιωτικά ντρόν κατασκευάζονται με ειδικέ προδιαγραφές και υψηλή κρυπτογράφηση που προσπαθεί να ελεγχιστοποιήσει στο βαθμό του δυνατού οποιαδήποτε τις πιθανότητες επίθεσης ή διείσδυσης αν θέλετε από τον εχθρό. Μπορώ τώρα εγώ να καθίσω σε αυτή τη θέση και να σας πω ότι 100% δεν υφίστανται παρεμβολές. Όχι, δεν μπορώ. Είναι αποτελεσματικά, είναι αποτελεσματική η προστασία και αν δει κανεί τα αριθμητικά στοιχεία πόσοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δουλεύουν με ντρόουν, Και αν δει κανεί το γεγονό ότι εξ όσων γνωρίζω δεν έχει υπάρξει κυβερνοεπίθεση τέτοιου είδου, όλα αυτά συντείνουν προ το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε. Ευχαριστώ. Και εγώ θα μπορούσα να σας δώσω παράδειγμα το RQ170, RQ170, μια πολύ προηγμένη τεχνολογία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπεσε στο Ιράν, δεν καταστράφηκε Ο πρώην πρόεδρος ζήτησε να του επιστραφεί και περιμένει ακόμα. Και το Ιράν κατάφερε να διεισδύσει στην τράπεζα δεδομένων αυτού του ντρόουν και απελευθέρωσαν και δημοσίευσαν ορισμένα βίντεο που έδειχναν το ντρόουν να πηγαίνει στον αεροπορικό διάδρομο μιας άλλης χώρας καθοδόν προς το Ιράν. Αυτά δηλαδή πρέπει κανείς να τα έχει υπόψη όταν χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένη στρατιωτική τεχνολογία. Ότι δηλαδή μπορεί να πέσει στα χέρια του εχθρού τελικά και να στραφεί μπούμεραν και να χρησιμοποιηθεί από την άλλη πλευρά, από τον εχθρό που είναι κάποιο άλλο κράτος, κάποιο έθνος, κάποια τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό είναι πρόβλημα, ναι. Για παράδειγμα, δεν θέλει κανείς να βάλει ένα μηχανισμό αυτοκαταστροφής του οχήματος, γιατί εάν ο διάβλος για να δώσουμε εντολή να αυτοκαταστραφεί ε, υποστεί hacking, θα μπορεί να μπει ο επιτιθέμενος, ο εχθρός σε αυτό το διάβλο και να δώσει αυτό την εντολή και να μας αυτοκαταστραφούν όλα τα οχήματα, τα αεροσκάφη, τα μη επανδρομένα που έχουμε. Σε πολλές περιπτώσεις χάσαμε UAV πάνω από το Λίβανο και επιτεθήκαμε σε αυτά τα επανδρομένα, μη επανδρομένα αεροσκάφη και τα καταστρέψαμε, τα δικά μας. Γιατί θελήσαμε να τα καταστρέψουμε και να προλάβουμε να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού, της Χεσμπολά ή του οποιοδήποτε άλλου. Αλλά δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε συνέχεια. Πολύ συχνά ένα ντρόν πέφτει στη θάλασσα και εξεβράζεται στη στεριά. Αυτό συνέβη για παράδειγμα πριν από ένα χρόνο. Πρέπει να τα ξέρουμε αυτά, να τα λαμβάνουμε υπόψη. Και πρέπει κανείς και να ρισκάρει. Υπάρχουν κάποιες πιθανότητες. Και εγώ θα ήθελα κάτι να συμπληρώσω, λέει ο κύριος Μάρεϊ. Το παράδειγμα του RQ170 είναι πολύ ενδιαφέρον. Να σας πω ότι όταν κάτι έχει προσγειωθεί, εν πάση προσεδαφιστεί και το παίρνουν οι εχθροί, το πάνε στο εργαστήριο και βάζουν τους επιστήμονες και ειδικού να το κοιτάνε και να το εξετάζουν, αυτό είναι κάτι το πολύ διαφορετικό από ένα ντρόν που πετάει και που προσπαθεί κανείς από το εργαστήριό του να το ελέγξει ή να, να κάνει hacking και να σπάσει την κρυπτογράφηση. Δηλαδή διαφορετικές μεθόδους ακολουθεί στη μία και στην άλλη ε, κατεύθυνση, στη μία και στην άλλη οπτική. Επίσης πολλά έθνη στο ΝΑΤΟ, όπως το Ισραήλ, έχουν χάσει μη επανδρομένα αεροσκάφη, έχουν χάσει drone, αλλά αυτό δεν οφείλεται στην κρυπτογράφηση και στην κυβερνοεπίθεση. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι λόγοι και εγώ εργάζομαι στις Βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις και έχω πάει στο Αφγανιστάν. Στην έρημο είχαμε πολλές απώλειες και τελικά στείλαμε ροσκάφη να τα καταστρέψουν τα ντρόν τα οποία είχαν καταπέσει όχι γιατί είχαν υποστεί θύμα, είχαν πέσει θύματα κυβερνοεπιθέσεων, αλλά γιατί είχαν κάποια δυσλειτουργία και χάλασε το μηχάνημα και έπεσε το ντρόν. Υπάρχει διαφορά δηλαδή και πρέπει να την τονίσουμε. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ε, υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά προβλήματα και υπάρχει και μία ευρή αναζήτηση να βρούμε τις απαραίτητες απαντήσεις. Κλείνει λοιπόν αυτό το πάνελ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες και θα ήθελα να δώσω το λόγο στις 11 όμως ε, στον κύριο Γκάλα που θα προεδρεύσει. Uh, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θα ξεκινήσουμε. Έτοιμοι να απογειωθούμε. Πάμε στο σημείο υπερθμών 9 τη ημερήσια διάταξης, ανταλλαγή απόψεων των Hans Peter Bartels, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικό εντεταλμένο ε, των ενόπλων δυνάμεων και των Ρενιέ Φαντζίτφεν, ο οποίος είναι ο εθνικό διαμεσολαβητής των ε, κάτω χρόνων της Ολλανδίας. Σας καλωσορίζουμε θερμά και Επειδή έχω αυτά που πρέπει να πω στα αγγλικά, ε, θα τα διαβάσω στα αγγλικά. Για όλα τα κοινοβούλια η εύρυθμη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων και η ευημερία των ανθρώπων που φορούν ε, στρατιωτική στολή είναι κάτι που πρέπει να είναι πολύ σημαντικό. Ε, πάρα πολλοί από τους στρατιώτες μας αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο εξωτερικό και συμμετέχουν σε ε, διάφορες επιχειρήσεις όπως ε, στο Trident ε, Juncture. Οι στρατιώτες οι οποίοι έχουν υπηρετήσει πολλές φορές τραυματίζονται, πεθαίνουν, πρέπει λοιπόν να είναι σωστά εξεπλισμένοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει όλοι. Καλούνται να αντιμετωπίσουν προβλήματα που έχουν σχέση με τη φύση, με το κλίμα, με το κρύο, με τις ε, τροπικές θερμοκρασίες ε, πρέπει να προσαρμόσουν τα καθήκοντά τους σε αστικό περιβάλλον και σε διάφορες περιοχές, σε λαούς, σε διάφορες γλώσσες. Καλούνται να ανταπεξέλθουν ε, σε αυτά το που έχουν δει, ζήσει, βιώσει με τα τραύματά τους, αλλά παρόλα αυτά όμως πρέπει να παραμένουν παράδειγμα υποδειγματική όσον αφορά τη συμπεριφορά τους και τη γενικότερη παρουσία τους. Αυτά λοιπόν ε, τους δημιουργούν στρες και μόνο αυτό αλλά και πολλά άλλα. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε στρατιωτικός πρώτα απ' όλα είναι άνθρωπος και πολίτης, ένας πολίτης ε, με στρατιωτική στολή. Οι Εθνικοί Επίτροποι και οι διαμεσολαβητές βρίσκονται και υπάρχουν ακριβώς αυτό για να μας υπενθυμίζουν ότι πρέπει να εισακούνται οι φωνές των στρατιωτικών. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τώρα τον κύριο Μπάρτελς να λάβει το λόγο και μετά θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Φαν Σούτφεν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γκάλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση ε, σε αυτή την ευρωπαϊκή θα την αποκαλούσα συνεδρίαση το δικό μου το αξίωμα, η δική μου θέση του εντεταλμένου για τις ένοπλες δυνάμεις, αυτό είναι κάτι το πολύ γερμανικό, ένα καθαρά γερμανικό, ένας γερμανικός θεσμός. Συστήθηκε όταν αποφασίστηκε η δυνατότητα της Δυτικής Γερμανίας να επανεξοπλίζεται. Και αυτό έγινε 10 χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν αμφισβητούμενο το κατά πόσο η Γερμανία θα έχει το δικαίωμα να εξοπλίζεται, να έχει στρατιώτες και θα γνωρίζετε φαντάζομαι ότι πολλοί θεωρούσαν ότι ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει γερμανικός στρατός και αν υπάρχουν γερμανοί στρατιώτες αυτοί θα πρέπει να αποσπώνται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Άμυνα. Η Γερμανία τότε ε, κύρωσε τις σχετικές συνθήκες, συμφώνησαν το Κοινοβούλιο και η κυβέρνηση. Τελικά όμως η Εθνική Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας ε, διαφώνησε και για το λόγο αυτό δεν υπήρξε Ευρωπαϊκό στρατός, άρα δηλαδή θα έπρεπε να σταθούν οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις. Για τους δημοκράτες στο Bundestag, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, κατέστη απόλυτα σαφές ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένας νέος στρατός. Καμία σχέση ούτε με το Reich, ούτε με το, τις παλαιότερες ένοπλες δυνάμεις. Μία πλήρης νέα σύσταση από το μηδέν. Και αυτή θα πρέπει να είναι ένας, ε, μια, θα πρέπει να είναι ένας στρατός που θα ελέγχεται από το Κοινοβούλιο, όχι από την εκτελεστική εξουσία. Αυτή η επανασύσταση του στρατού θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις σε τελική ανάλυση να εξαρτάται από την απόφαση του Κοινοβουλίου. Ακόμα και σε περίπτωση άμυνας, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και το Bundestag και το Bundesrat είναι εκείνα τα οποία έχουν την τελική λέξη. Και στο Σύνταγμά μας αναφέρεται ότι αν τελικά το Bundestag δεν μπορεί πλέον να συνέλθει και μπορείτε να φανταστείτε το τι σημαίνει αυτό, τι είχαν κατά νου όταν ε, έκαναν αυτή τη διατύπωση, τότε θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος έκτακτου κοινοβουλίου, ένα μίνι κοινοβούλιο, το οποίο θα λάβει την τελική απόφαση. Δηλαδή, και πάλι αναφέρεται ότι θα πρέπει να λαμβάνεται μια κοινοβουλευτική απόφαση για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο στρατός τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, κάτι το οποίο βιώσαμε ε, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Για κάθε περίπτωση που συμμετέχουν Γερμανοί στρατιώτες, καλείται να αποφασίσει το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Κατόπιν, το Σύνταγμα ε, έχει προβλέψει δύο ειδικού θεσμούς για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας το 45α του συντάγματος, εκεί προβλέπεται ε, Επιτροπή Άμυνας. Υπάρχει σε όλες τις χώρες, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ίσως είναι υποεπιτροπή, αλλά σε κανονικά κοινοβούλια είναι κανονική επιτροπή. Άρα πρέπει να υπάρχει Επιτροπή Άμυνας. Δεν μπορεί δηλαδή να πει κανείς έχουμε μια επιτροπή για άμυνα, αθλητισμό και πολιτισμό. Όχι, αμυγός ε, ε, αμυντική επιτροπή. Και αυτή η Επιτροπή έχει δικαιώματα με βάση το άρθρο που σας είπα 45α. Στο άρθρο 45β του συντάγματός μας αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας εντεταλμένος για θέματα ενόπλων δυνάμεων. Αυτόν θα, τον ορίζει το Κοινοβούλιο και ε, ο εντεταλμένος αυτός έχει το μόνιμο έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων και είναι και ο συνομιλητής για κάθε ένα και μεμονωμένο στρατιώτη, οποτεδήποτε ο στρατιώτης αυτός αισθάνεται ότι παραβιάζονται τα στρατιωτικά και τα ατομικά του δικαιώματα. Τότε ο στρατιώτης ε, μπορεί να απευθυνθεί στο Κοινοβούλιο Άρα δηλαδή κάθε στρατιώτης ανεξάρτητα από την υπηρεσιακή οδό μπορεί να απευθυνθεί στον εντεταλμένο ε, στρατιωτικών δυνάμεων. Αρχικά βέβαια ε, η σκέψη ήταν ότι με τον τρόπο αυτό ε, θα πρέπει να εμποδιστούν οι παλιές μέθοδοι της Wehrmacht γιατί η Wehrmacht είχε συσταθεί από αξιωματικούς και από στρατιωτικούς οι οποίοι είχαν υπηρετήσει. Στην αρχή έτσι και αλλιώ δεν υπήρχε και κανένα άλλο. Μετά όμω θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν νέε αρχέ, να ισχύσουν νέε εκπαιδευτικέ αρχέ. Έχουμε λοιπόν στη Γερμανία νέε αρχέ, οι οποίε για μα αποκαλούνται εσωτερική καθοδήγηση. Και αυτό συμπληρώνει την γνωστή εξωτερική καθοδήγηση που αφορά τις ε, εντολές ε, και την ε, υπακοή. Όποιος λοιπόν θέλει να ε, τις αγνοήσει αυτές τις δύο αρχές μπορεί να ε, καταδικαστεί σε θάνατο. Η Bundeswehr λέει ότι εκτός από αυτές τις δύο αρχές της εντολής και της υπακοής μπορεί να υπάρχει και κάτι παραπάνω, είναι η συνείδηση. Η συνείδηση και οι αρχές ε, τις οποίες πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του. Αρχές λοιπόν για το καλό, το αγαθό και το κακό, για το σωστό και το λάθος, για το δίκαιο και το άδικο. Κάθε μεμονωμένο στρατιώτης πρέπει να ε, εμφορείται από αυτές τις αρχές και αν παραβιάζονται αυτές οι αρχές δεν πρέπει να εκτελεί εντολές. Στο Σύνταγμα της Γερμανίας υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες ενδιαφέρουσες απόψεις και διατυπώσεις που έχουν βέβαια σχέση και με το παρελθόν. Μία εξ αυτών βρίσκεται στο 24 και το άρθρο 24 δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Για να τροποποιηθεί το άρθρο 24 πρέπει να καταργηθεί το Σύνταγμα. Το άρθρο αυτό είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του Συντάγματος και εκεί αναφέρεται ότι οποιοδήποτε προσπαθήσει να παραβιάσει αυτόν τον ε, δημοκρατικό έλεγχο, ε, στην περίπτωση αυτή δικαιολογείται η αντίσταση. Και γιατί αναφέρεται αυτό, γιατί υπήρξε μια τέτοια κατάσταση πριν από κάποια χρόνια, Το 1944 στρατιώτες της ε, Wehrmacht, τότε του στρατού, παραβίασαν τον όρκο τους ε, στον Χίτλερ, παραβίασαν τις εντολές και την υπακοή και προσπάθησαν ε, να ανατρέψουν το καθεστώς με πραξικόπημα. Και που βασίστηκαν μόνο στη συνείδησή τους, στα δικά τους τα κριτήρια, μέτρα και σταθμά για το αγαθό και το κακό και ήταν λοιπόν αναγκασμένοι να πράξουν με βάση το σύνταγμα που ίσχυε τότε λάθος, αλλά με βάση που ίδιοι, αυτό που πίστευαν οι ίδιοι το σωστό. Και γι' αυτό σκέφτηκαν οι Γερμανοί, ας το γράψουμε και αυτό στο σύνταγμα, ότι είναι σημαντικό να διατηρούμε τις, ε, τα δικά μας, ε, τα ανθρώπινα κριτήρια, τα δημοκρατικά κριτήρια. Όλοι οι στρατιώτες πρέπει να το έχουν αυτό στη Γερμανία, όλοι οι στρατιώτες πρέπει να θέλουν να υπερασπιστούν τη δημοκρατία. Αν δεν το θέλουν, δεν μπορούν να είναι στρατιώτες στρατιώτες των ε, ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας. Πρέπει να έχουν κατά νου την ελευθερία, αλλιώς δεν μπορούν να είναι στρατιώτες στη Γερμανία. Όχι μόνο να αγωνίζονται και να μάχονται, αλλά να γνωρίζουν και γιατί πράγμα ακριβώ μάχονται. Αυτό είναι ένα από τα κριτήρια του νέου στρατού μετά από τι εμπειρίε που κάναμε ε, με του δύο προηγούμενου στρατού. Και η Reichsmacht ε, και αυτό δεν ήταν καλός ε, στρατός ε, ε, και αυτός είδαμε ότι δεν αποδείχθηκε χρήσιμος μέσα στις ιστορικές εξελίξεις. Έχουμε λοιπόν μια μακρά εμπειρία και καταλήξαμε στο ότι χρειαζόμαστε κοινοβουλευτικό έλεγχο του συνόλου των ενόπλων δυνάμεων. Όλοι οι στρατιώτες θα πρέπει να έχουν κατά νου τα δικά τους ακριτήρια, να μπορούν να απευθύνονται στο Κοινοβούλιο. Αρχικά λοιπόν επρόκειτο καθαρά για θέματα ε, μιλιταρισμού και παράδοσης της Wehrmacht. Δηλαδή αυτή η νέα αρχή της εσωτερικής καθοδήγησης κατά πόσον μπορεί αυτή να εφαρμοστεί. Και με αυτό είχαν προβλήματα και αναγκάστηκαν να αγωνιστούν οι προκάτοχοί μου και ο πρώτος και ο δεύτερος και αναγκάστηκαν να παρατηθούν στον αγώνα με την κυβέρνηση, με τους αξιωματικούς, με το κοινοβούλιο παρεπιπτόντος και οι δύο, ο ένας ε, ήταν πρώην ε, στρατηγός, ο άλλος ήταν ναύαρχος και οι δύο με το κλασικό βιογραφικό που υπήρχε τότε στη Γερμανία. Ε, αυτοί λοιπόν είχαν μάθει με το παλιό καθεστώς, θέλησαν όμως να εργαστούν με το καινούριο. Οι δύο λοιπόν προκάτοχοί μου ήταν εκείνοι οι οποίοι υπερασπίστηκαν αυτή την αρχή της εσωτερικής καθοδήγησης μέχρι και την παρέτησή τους. Ο δεύτερος μάλιστα δημοσίευσε τις απόψεις του στον τύπο γιατί εντωμεταξύ δεν μπορούσε τότε να μιλήσει στο κοινοβούλιο. Ε, εγώ μπορώ να απευθυνθώ στο Κοινοβουλίο. Ήμουν 17 χρόνια βουλευτή, ε, τώρα δεν είμαι πια βουλευτή. Δεν είμαι βέβαια ούτε υπάλληλο. Είμαι κάτι στη μέση είναι μια sui generis, ένα sui generis ε, θεσμός, όπως λένε και οι συνταγματολόγοι, και έχω το δικαίωμα να λαμβάνω το λόγο. Μία φορά το χρόνο ε, καταρτίζω μια έκθεση για το Κοινοβούλιο, 100 σελίδων, και εκεί η δική μου υπηρεσία που έχω περίπου 50 συνεργάτες ε, και εγώ ε, αναφέρουμε ποιες είναι οι παρατηρήσεις μας, ε, ποια είναι τα κακό σκήμενα, τι αναφέρουν οι στρατιώτες, τι πρέπει να βελτιωθεί. Αυτή λοιπόν την έκθεση την παραδίδουμε στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο οποίος την καταθέτει στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Μετά η έκθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή Άμυνας που αυτή απευθύνεται στην γερμανική κυβέρνηση η οποία και τοποθετείται και μετά ε, υπάρχει μια δεύτερη ανάγνωση στο Γερμανικό Κοινοβούλιο όπου πλέον ε, γίνονται διαβουλεύσεις για την έκθεση της προηγούμενης χρονιάς. Πρέπει να σας πω ότι εντωμεταξύ δεν πρόκειται κατά κύριο λόγο ε, για το κατά πόσον πρέπει να αγωνιστούμε κατά του μιλιταρισμού ή όχι. Η κυβέρνηση που έχουμε και ο στρατός που έχουμε σήμερα είναι ένας δημοκρατικός στρατός ε, ο οποίος λειτουργεί με βάση δημοκρατικές αρχές δηλαδή όλοι οι στρατιώτες θα πρέπει να είναι δημοκράτες ε, και όλοι οι στρατιώτες έχουν δικαίωμα σε πολιτική, ιστορική, ηθική εκπαίδευση. Υπάρχει δηλαδή και διδασκαλία στο στρατό Όλα αυτά συνδεμένα πάντα με την εσωτερική καθοδήγηση. Όλοι οι στρατιώτες έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε. Έχουμε αρκετούς ε, στρατιώτες και στρατευμένους ε, στο Κοινοβούλιο. Βεβαίως όσο υπηρετούν ε, είναι αποσπασμένοι. Μπορούν όμως αργότερα αν θέλουν να επανέλθουν. Έχουμε πάρα πολλούς στρατευμένους που επίσης εργάζονται στα τοπικά κοινοβούλια. Οι στρατιώτες και οι στρατευμένοι μπορούν να είναι και μέλη συνδικάτων. Ε, οι στρατιωτικοί έχουν μάλιστα και ένα συνδικαλιστικό όργανο με 200 μέλη που μιλάνε συνεχώς για το τι πρέπει να αλλάξει στο γερμανικό στρατό. Αναζητούν λύσεις. Οι στρατιώτες ε, ε, έχουμε τους εκπροσώπους τους και έχουμε ε, εκείνους όλους που τους εκπροσωπούν. Οι στρατευμένοι έχουν επίσης ε, και το δικαίωμα να απευθυνθούν στον εντεταλμένο, αν πρόκειται για θέματα στρατού. Αν είναι θέματα άλλα που τους απασχολούν, παραδείγματος χάρη για την σύνταξή τους ή οτιδήποτε, θα απευθυνθούν στην Επιτροπή Αναφορών. Αλλά αν αυτά που θέλουν να θίξουν στρατιωτικά θέματα, θα έρθουν σε μένα. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα δικαιώματα εγώ κάθε χρόνο έχω περίπου 2.500 ε, αναποφορές ε, από 1.800 ε, περίπου στρατευμένους, δηλαδή Όλοι ε, κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματός τους ε, και οποτεδήποτε ε, αναφέρονται περιπτώσεις εκφοβισμού σεξουαλικών παρενοχλήσεων ή άλλων προβλημάτων γιατί παραδείγματος χάρη υπήρξαν και προβλήματα πέρυσι όπου κάποιοι πέθαναν στη βασική εκπαίδευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρεμβαίνουμε εμείς και παρακολουθούμε την υπόθεση και σε τελική ανάλυση μιλάμε για 4.500 αναφορές το χρόνο που παρακολουθεί η υπηρεσία μου και όπου όταν πρόκειται για μεμονωμένους στρατιώτες ε, πολύ συχνά ε, μπορούμε να επιτύχουμε το θέμα να λυθεί προς όφελός τους. Και αυτό φτάνει μέχρι ε, και το τι πρέπει να γίνει ε, με τη μεταφορά σε μάχες, σε θέατρα μάχης. Ε, Παραδείγματο χάρη το πώ θα μεταφερθούν οι στρατιώτε σε αυτά τα θέατρα πολέμου και όχι να αναγκασμένοι να περιμένουν ε, πότε θα έρθει η κατάλληλη πτήση. Μην ξεχνάτε ότι και οι στρατευμένοι έχουν οικογένειε και είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να συνδυάσουν και τον οικογενειακό του ε, βίο, την οικογενειακή του ζωή. Έχουμε ανθρώπου ε, οι οποίοι πολλέ φορέ είναι άνω τη ηλικία των 30-35 ετών. Αυτοί μεταξύ έχουν τη δική του οικογένεια και οι άνθρωποι αυτοί θέλουν και αυτοί να δουν τα παιδιά τους και οι άνδρες και οι γυναίκες. Σήμερα λοιπόν είναι άλλα θέματα που μας απασχολούν. Είναι ο εξοπλισμός, είναι ο συμβιβασμό της υπηρεσίας με την οικογένεια. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία πολλές φορές θίγονται σε μένα και που πολλές φορές βέβαια έχουν και άμεση σχέση με τα βασικά δικαιώματα των στρατευμένων. Εάν οι στρατευμένοι ε, δεν ε, έχουν ε, εκπαιδευτεί σωστά, τότε δεν μπορούν να είναι και επιτυχημένοι στην, ε, την ώρα που καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Άρα δηλαδή η εκπαίδευση και ο σωστός εξοπλισμός είναι κάτι απολύτως απαραίτητο σήμερα στη Γερμανία. Ε, μέχρι το 2014 ο δικός μας ο στρατός ε, χρησιμοποιεί το μόνο εκτός της Γερμανίας. Ε, την εποχή του ψυχρού πολέμου υπήρχε μόνο μία περίπτωση της συλλογικής άμυνας. Τώρα όμως υπάρχουν και τα δύο. Έχουμε την ανάπτυξη στρατευμένων εκτός Γερμανίας, αλλά αυτό που είναι κάτι το καινούριο το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι οι στρατιώτες μας μπορούν πλέον να συμμετέχουν στην συλλογική άμυνα, όχι για γιατί έχουμε ψυχρό πόλεμο, αλλά διότι και πάλι κρίνεται απαραίτητο να συμμετέχουν οι στρατιώτες σε ένα ελάχιστο εκφοβισμού. Υπάρχουν βέβαια πολλά κενά στο προσωπικό, ε, πάρα πολλοί ε, καλούνται να καλύπτουν θέσεις που ε, για μια συγκεκριμένη στιγμή χειρεύουν. Επίσης το υλικό και ο εξοπλισμός πολλές φορές δανείζεται αυτός, ε, τα λεξίσφαιρα γυλαίκα, αυτά πολλές φορές πηγαίνουν και έρχονται. Αυτό βέβαια δεν είναι και καλό, δεν είναι σωστό. Λείπει εξοπλισμός, λείπει η εκπαίδευση. Αυτά είναι τα θέματα για τα οποία διαμαρτύρονται οι στρατιώτες. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια διαφορετική κατάσταση όπως πριν από 16 χρόνια όταν πρωτοσυστήθηκε η δική μας υπηρεσία. Σήμερα η δουλειά είναι τελείως διαφορετική. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπάρτελς για την εικόνα που μας παρουσιάσατε που πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Βέβαια σαφώς και υπάρχει μια ιδιομορφία στην περίπτωση της Γερμανίας λόγω της προϊστορίας. Αλλά οι στρατευμένοι ανεξάρτητα που υπηρετούν και σε ποιο στρατό νομίζω ότι ε, παντού αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Τίτε λοιπόν το ερώτημα ποιο δρόμο μπορούν να ακολουθήσουν οι στρατευμένοι έτσι ώστε να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Να καλωσορίσουμε θερμά τον ε, κύριο Βαν Σίτφεν από τις 100 χώρες. Έχετε και άλλους ε, πελάτες βέβαια υπό την ιδιότητά της, αλλά, σας, συγγνώμη, αλλά σήμερα θα μας μιλήσετε για την ε, κατάσταση της 100 ε, χώρες ε, σε σχέση με τους ενστόλους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας πω δύο λόγια για το έργο επειδή είμαι βετεράνος σε αυτόν τον τομέα πριν από 35 χρόνια συστάθηκε η θέση του Ολλανδικού Συνηγόρου Ναι, συνεχίζω. Πριν από 35 χρόνια λοιπόν συστάθηκε αυτή η θέση που εξετάζει ε, τα παράπονα και τις καταγγελίες των πολιτών σε όλα τα επίπεδα και σε εθνικό και σε περιφερειακό και σε τοπικό, σε όλους ε, τους ε, τομείς όπου έχουμε δημόσια δράση, ε, αστυνομία, επιδόματα, Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν στο δημόσιο βίο έχει να κάνει με τις δικές μας αρμοδιότητες. Το 2014 υιοθετήθηκε ένας ε, τέτοιος ε, νόμος ε, στις κάτω χώρες για τους βετεράνους πιο συγκεκριμένα. για στρατιώτες που έχουν συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις ή και ειρηνευτικές αποστολές και θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο να δώσουμε ιδιαίτερη μέρημνα και φροντίδα σε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα πλέον που έχει συσταθεί για την σωστή υποδοχή και αντιμετώπιση των βετεράνων και προέκυψε ότι πρέπει να υπάρχει ένας εξωτερικός ε, συνήγορος του πολίτη, αν θέλετε, για την, ή των βετεράνων εμπροκειμένο, σε εθνικό επίπεδο, ε, που έχει πολύ καλή εμπειρία ε, στην επεξεργασία τέτοιων παραπώνων. Επομένως, πλέον ο συνήγορος του πολίτη έχει γίνει και συνήγορος των βετεράνων. Προηγουμένω πρόκειται για άτομα τα οποία είχαν πολεμήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε πολλά ερωτήματα που προέκυψαν μετά από την ε, ε, πολεμική αυτή σύραξη. και από τις 100 χώρες, από την Ολλανδική Ινδία, την Κορέα. Είναι ακόμα εν ζωή πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους και απευθύνονται στον ε, ε, συνήγορο των βετεράνων. Και οι και πολλέ άλλε ε, χώρες ε, έχουν συμμετάσχει σε ειρηνευτικέ αποστολές και συμμετικές επιχειρήσεις. Γι' αυτό έχουμε ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει στο Λίβανο, στο Κοσμοπέδιο, το Αφγανιστάν, το Μαλί. Εκεί δημιουργούνται αυτή τη στιγμή, α το πούμε έτσι, οι βετεράνοι. Και πρόκειται για νέου ανθρώπου, ενεργού στο πεδίο γιατί όταν λέμε βετεράνους συνήθως ε, σκεφτόμαστε μόνο τους ε, ε, αλλά όχι εδώ πρόκειται και για νέους ανθρώπους, ε, τριαντάριδες, άνδρες, γυναίκες, με, μια σειρά προβλήματα. Και βλέπουμε ότι για αυτούς είναι πολύ σημαντικός αυτός ο θεσμός ε, του συνηγόρου των βετεράνων. Κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός ε, των αιτήσεων και καταγγελίων που λαμβάνουμε. Ε, Ιδίω τα τελευταία χρόνια έχουμε λάβει πολλαπλάσιες αιτήσει και αναφορές. Και πρέπει ε, να σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι πρόκειται για ανθρώπους που υπηρέτησαν στο Αφγανιστάν, έπεσαν πάνω σε ενέδρα ή βόμβα ε, και ότι μετά είναι δύσκολη η περίθαλψή τους, η επανένταξή τους, ε, τα εισοδήματά τους πλέον, τα κοινωνικά επιδόματα, η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Για μας μαζί με το συνεργάτη μου που με συνοδεύει σήμερα σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πολύ έντονες επαφές ε, και σχέσεις με τους βετεράνου. Εμείς συμμετέχουμε σε όλα τα πεδία όπου συγκεντρώνονται οι βετεράνοι και έτσι προσπαθούμε να ε, προαγάγουμε την οργάνωσή τους ε, για να έχουν την καλύτερη δυνατή ζωή. Ε, δεν εξετάζουμε μόνο μεμονωμένες αιτήσει και αναφορές, μπορούμε να κάνουμε και έρευνες με δική μας πρωτοβουλία. Όταν λοιπόν λαμβάνουμε ενδείξει ότι κάπου κάτι δεν πάει καλά, μπορούμε, κάτι το οποίο εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό, να αναλάβουμε δράση ε, από μόνοι μα. Και θεωρώ ότι πολύ σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα ε, οι ίδιοι άνθρωποι να μπορούν να καταγγέλουν τα κακό κείμενα στη χώρα τους και αυτό αρχίζει να αυξάνεται και το έχουμε συμπεριλάβει εμείς στην έκθεσή μας να υπάρχει καλύτερη λοιπόν ε, επεξεργασία των ε, αναφορών, γιατί μέχρι τώρα ήταν ε, ελλειπής. Στη συνέχεια με τον Υπουργό συζητήσαμε και είπαμε ότι συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να μεριμνούμε για το ίδιο το σύστημα επεξεργασίας αναφορών και καταγγελιών. Πρέπει να βελτιωθεί. Στον αναδικό στρατό είναι μεγάλο το πρόβλημα και σε ό,τι αφορά την, τον εκφοβισμό, σεξουαλική και σεξουαλικός εκφοβισμός, απειλές, ε, συστήματα ναρκωτικών. Είναι πολύ δύσκολο για τους ενστόλους να τα καταγγείλουν όλα αυτά. Γι' αυτό είμαστε εμείς εκεί λοιπόν. Ε, θα μείνω εδώ. Έχουμε στείλει ένα έγγραφο, μια έκθεση ε, όπου παρουσιάζουμε τις δραστηριότητές μας. Μπορείτε να τα βρείτε λοιπόν όλα αυτά και εκεί και με χαρά να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις vielen Dank, äh, Και εμεί ευχαριστούμε πολύ. Αυτά που μας είπατε ε, κατέδειξαν ότι η δομή είναι τελείω διαφορετική. Για μας λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ ενδιαφέρον το να βλέπουμε το πώς ακριβώς ε, μπορεί κανείς ε, να διατυπώσει τα συμφέροντα των ε, στρατευμένων, ε, τι είδου ε, προσεγγίσεις υπάρχουν, διαφορετικές προσεγγίσεις. Έχουμε επαφή και με την Euromill, τον οργανισμό που εκπροσωπεί τους στρατευμένους. Τα πράγματα πραγματικά είναι πολύ διαφορετικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να τεθεί το ερώτημα τελικά όταν είμαστε καθοδόν. Ισχύουν κοινέ διατάξεις για όλους τους στρατιώτες και στο μέλλον οι στρατευμένοι πού θα πρέπει να απευθύνονται όταν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο ε, κατά διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος ε, στην ομάδα εργασία Καγκουρού που έχουμε συστήσει. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω τον γύρο των ερωτήσεων ε, παρακαλώ, οι συνάδελφοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις. Ο κύριος Έιλαρ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας καλωσορίσω εκ μέρους του ΕΛΚ. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Ε, καταρχήν προς τον κύριο Μπάρτελς. Το Σαββατοκύριακο η Καγκελάριος και ο πρόεδρος Μακρόν θέλησαν ε, κάπως να προωθήσουν λιγάκι αυτή την ιδέα του Ευρωπαϊκού στρατού. Οι εθνικοί στρατοί εδώ και χρόνια και των δύο χωρών συμμετέχουν ε, εδώ και αρκετές δεκαετίες ε, στο ΝΑΤΟ. Βεβαίως είναι διαφορετικά οργανωμένοι οι δύο αυτοί στρατοί. Στο θέμα όμως του Ευρωπαϊκού στρατού τίθεται και το ερώτημα του πώς γίνεται η διαχείριση των ε, στρατών αυτών στις δύο χώρες. Στη Γαλλία έχουμε ένα τελείως διαφορετικό σενάριο ε, που ισχύει παραδείγματο χάρη για τη λεγιώνα των ξένων, το πώς ε, αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται αυτή η λεγιώνα, αλλά υπάρχουν και άλλες μονάδες, γαλλικές μονάδες, οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν σε διενέξεις με τρίτες χώρες. Αυτή είναι η οργάνωση, η δομή που υπάρχει στη Γαλλία. Και θέλω να ρωτήσω, για να γίνει έτσι κάπως πιο κατανοητό το θέμα της ε, διαχείρισης ε, στρατών και τρόπου ε, διακυβέρνησης τους, υπάρχουν κάποιες απόψεις ε, οι οποίες να αφορούν, ε, παραδείγματος χάνει, τη χρήση αυτών των στρατευμάτων για ασύμετρες ε, επιθέσεις, για μικτές αποστολές, από κοινού με αστυνομικές δυνάμεις. Εσείς που είστε ε, τι ακριβώς κάνετε, ασχολείστε μόνο με το γερμανικό στρατό, μόνο με την Bundeswehr ή υπάρχει και ένας ευρωπαϊκός διάλογος. Γιατί, παραδείγματος χάρη, στην αντιμετώπιση τρομοκρατίας σε τρίτες χώρες, προφανώς εκεί υπάρχουν ε, κοινά επιτελεία και υπάρχουν ε, κοινά σχήματα ανάπτυξης επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο να ακούσουμε και να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται για να προστατευτούν τα δικαιώματα των στρατιωτών μας που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. Κατανοώ τους το υπόβαθρο της γερμανικής Wehrmacht. Λόγω του παρελθόντος της. Ωστόσο, τα δικαιώματα αυτά ισχύουν πλήρως για τις ένοπλες δυνάμεις εν καιρό ειρήνης. Τι συμβαίνει όμως σε κατεξαίρεση περιστάσεις, σε εξαιρετικές συνθήκες, σε περίπτωση επίθεσης σε περίπτωση ανάγκης να αντιταχθεί κανείς στον επιτιθέμενο και στον κατακτητή. Διότι ναι, για να αποφύγουμε τις πρακτικές του παρελθόντος, δηλαδή οι στρατιώτες να υπακούν τις διαταγές όποιες και να είναι, ακόμα και αν είναι ποινικό κολάσι θα περίμενε κανείς να αυτό να συμβαίνει σε καταστάσεις δικτατορίας. Όμως, είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε πράγματι να δοθούν εγκληματικές εντολές από δημοκρατική ηγεσία σε δημοκρατικά καθεστώτα. Και όσοι μπαίνουν στο στρατό πρέπει να το γνωρίζουν πολύ καλά. Να γνωρίζουν πολύ καλά πού πηγαίνουν, σε ποιο σύστημα προσχωρούν, Μπορείτε να φανταστείτε εν καιρό πολέμου και εν καιρό κρίσεις και ειρήνες να ε, προβάλλουν οι στρατιώτες την ατομική του συνείδηση εδώ και εκεί. Το οποίο είναι απόλυτο κατανοητό σε μια ευρία κλίμακα, αλλά πώς θα ταιριάξει με αυτή την επίγουσα κατάσταση. Και εσείς μιλήσατε για δημοκράτες στρατιώτες με δημοκρατική νοοτροπία όταν στρατολογούνται. Η ερώτησή μου στην πράξη όμως είναι η εξής τα μέλη του ΑΕΦΔ ή νεοναζί μπορούν να μπουν στο γερμανικό στρατό. Ή μπορεί κανείς να αποβληθεί από το γερμανικό στρατό γιατί είναι ακροδεξιός ή έχει μη δημοκρατική, δημοκρατικό πολιτικό φρόνημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φρόιντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, ζητώ συγγνώμη καταρχήν γιατί καθυστέρησα να έρθω και ως εκ τούτου ε, δεν γνωρίζω ακριβώς ε, το τι είπατε. Δεν μπορώ δηλαδή να βασιστώ και να κάνω ρωτήσεις αυτά που είπατε. Όμως, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο συνάδελφός μου, ο Κρίστιαν Έιλερ. Και προσπαθώ και εγώ να διατυπώσω μία ερώτηση ε, που να ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση για να μην μου πείτε μετά εκτός θέματος. Θα ήθελα να μιλήσω για το αγαπημένο μου θέμα, το οποίο έμεσα έχει σχέση με αυτά τα οποία μάλλον αναφέρατε. Δηλαδή, θα ήθελα εγώ να κάνω ένα ερώτημα ε, σχετικά με την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική που δυστυχώς δεν υπάρχει κατ' εμέ. Το είπε και ο Κρίστιαν αυτό προηγουμένως. Έχω την εντύπωση ότι με αυτή την κοινή άμυνα των κοινό στρατό που προβάλλεται όλο και περισσότερο, κατ' ουσίαν τι συμβαίνει. Χρησιμοποιούμε ένα σχήμα προθύστερο. τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Θα ήταν πολύ πιο απλό να χαράξουμε μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, αυτή να προηγηθεί και μετά να ασχοληθούμε με ευρωπαϊκή κοινή αμυντική πολιτική. Και θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, δυστυχώς ε, μη πραγματοποιηθεί σαν κοινή εξωτερική πολιτική έναντι της Ρωσίας. Έχουμε τη Συμφωνία Μίνσκα 2 και εκεί τι έχουμε. Έχουμε δύο ευρωπαϊκά κράτη που εκπροσωπούν την Ευρώπη, αλλά δεν έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει το γεγονός ότι ε, Έχουμε στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 500 εκατομμύρια πολίτες. Είμαστε μια ισχυρή οικονομική δύναμη. Κατόπιν τούτου, ως τέτοια, θα μπορούσαμε να επιτύχουμε πολλά περισσότερα ε, στις σχέσεις μας με τη Ρωσία και κυρίως ε, όσον αφορά τα ε, τεκτενόμενα στην Ουκρανία. Πολύ περισσότερα από ό,τι τα έχουν επιτύχει τα δύο κράτη που μας εκπροσωπούν. Ερωτώ λοιπόν συγκεκριμένα, δεν πιστεύετε κι εσείς ότι θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο έτσι ώστε η Ευρώπη προς τα έξω να εμφανίζεται πιο ενωμένη όσον αφορά τη διπλωματία. Και εκεί που αποτυγχάνουν οι διπλωμάτες, εκεί πράγματι να μπορεί κανείς να εμφανίζεται με ε, κοινό ευρωπαϊκό στρατό και στρατιωτικά μέσα. Και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο ε, στους ε, δύο εισηγητές μας, πρώτα στον κύριο Μπάρτελς. Κύριε Έιλαρ, ε, αυτό που δείξατε εσείς πράγματι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και ένα θέμα που ακόμα δεν συζητιέται. Άρα δηλαδή Ας το ξαναπώ με σαφήνεια. Δεν μιλάμε για την εσωτερική διαχείριση του στρατού, αλλά τα δικαιώματα των στρατευμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποικίλουν πάρα πολύ. Στη Ρουμανία, παραδείγματο χάρη. Εκεί αυτά που είπα, δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεστε ή τον ένα οι στρατευμένοι μέλη συνδικάτων, αυτά δεν υπάρχουν. Σε εμά υπάρχουν, σα το εξήγησα. Τελείω διαφορετική εμπειρία στη Ρουμανία, άλλος πολιτισμός, άλλε. Ε, ε, ιστορικές ε, καταβολές. Ως εκ τούτου σας λέω, εμείς στη Γερμανία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχουν δημοκρατικά δικαιώματα για τους στρατευμένους. Και όπως τα αναφέρει το Σύνταγμα, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ καλό. Ως εκ τούτου, εγώ δεν είμαι αναγκασμένος να θεσπιστούν αυτά τα δικαιώματα, απλά αυτό που εγώ πρέπει να κάνω είναι να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα αυτά. Μόνο που στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδιώξουμε ένα είδος εναρμόνησης, αυτό που είπε και ο φίλος μας εδώ, να υπάρχουν κοινά στοιχεία. Βεβαίως και να υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική, αλλά για δέστε, εγώ ξεκίνησα με τα δικαιώματα των ε, στρατευμένων, με τα ατομικά τους δικαιώματα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, να δούμε τι δικαιώματα έχει ο κάθε ένας εξ αυτών, ε, τι δικαιώματα έχει και ως πολίτης. Ίσως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να επιληφθεί αυτού του θέματος να δρομολογήσει μια συζήτηση ανάμεσα στα διάφορα κράτη, γιατί όσον αφορά τα δικαιώματα των στρατευμένων, νομίζω ότι αυτό είναι καθαρά εθνικό ε, θέμα, εθνική αρμοδιότητα. Και βεβαίως αυτά ε, θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πλαίσιο, είναι πολύ βασικά, στο πλαίσιο μιας κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας, αν την επιθυμούμε αυτήν. Υπάρχει και το θέμα ε, του ε, γερμανικού στρατού εν καιρό που είναι δημοκρατικός στρατός, ευτυχώς θα έλεγα. Ευτυχώς εδώ και 60 χρόνια ο γερμανικός στρατός ε, έχει συνεισφέρει έτσι ώστε να μην υπάρξει πόλεμος. Το μεγάλο μας καθήκον ήταν να συμμετέχουμε σε επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες αλλά και οι Γάλλοι ε, ανέκαθεν ε, έβλεπαν το στρατό τελείως διαφορετικά. Δηλαδή είναι της άποψη ότι ο στρατός υπάρχει για να ε, μάχεται. Οι Γερμανοί τι λένε και πιστεύουν. Όχι, στρατός ποτέ να μην επεμβαίνει. Γιατί ε, αν είχαν συμμετάσχει μέχρι τώρα στρατιώτες σε κάποιες εμπόλεμες καταστάσεις, είχαμε καταλήξει και σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Σας λέω, οι Γερμανοί λένε ναι στρατός, αλλά ποτέ να μην επεμβαίνει. Οι Αγγλοσάξονες τα βλέπουν διαφορετικά. Δεν τι έγινε στα Φόρκλαντ, σε και αλλού. Εμείς έχουμε όλες αυτές τις δεσμεύσεις που υπάρχουν από το παρελθόν, αλλά έχουν και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι με τη Φραγκοφωνία, με την Κοινοπολιτεία. Τελείως διαφορετικές νοοτροπίες, τελείως διαφορετικοί πολιτισμοί. Ο γερμανικός στρατός ε, δεν έχει συσταθεί για να συμμετέχει σε μακρινές ε, ε, αποστολές, αλλά τώρα κάπως συμμετέχει στο Αφγανιστάν και αλλού και οι φίλοι μας όταν μας ρωτάνε τι γίνεται με τη συνεργασία, εγώ θα έλεγα η συνεργασία είναι καλή. Παραδείγματο χάνει στο Αφγανιστάν, οι Γερμανοί δεν, ήταν, δεν συμμετείχαν μόνο σε ήπια μέτρα, αλλά και σε ουσιαστικά μέτρα επίθεσης. Είχαμε τους Αμερικανούς, οι οποίοι στο Αφγανιστάν συμμετείχαν στις επιθέσεις και ε, στην περίπτωση αυτή, αν οι Γερμανοί έκαναν πίσω, νομίζω θα ε, καταλήγαμε σε αποτυχία. Και δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Άρα δηλαδή αυτό που πρέπει να συζητήσουμε και να καταλήξουμε είναι ποια στρατηγική είναι ελπιδοφόρα. Και εκτός από τα Βαλκάνια, όπου πράγματι η στρατιωτική επέμβαση ήταν επιτυχημένη, γιατί αυτό που μπορούσε να γίνει στα Βαλκάνια έγινε, τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει ε, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να κερδιθεί χρόνος για να υπάρξουν μη στρατιωτικές ε, εξελίξεις. Βέβαια, στο Αφγανιστάν αυτό δεν το καταφέραμε, ούτε και στη Λιβύη, ως εκ τούτου πρέπει να υπάρχει μία επιτυχημένη παρέμβαση. Σε δύσκολες καταστάσεις δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα. Ως εκ τούτου πρέπει να συζητήσουμε για το πώς μπορούν να στέφονται από επιτυχία οι αποστολές. Ε, εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Βέβαια και οι Βρετανοί και οι Γάλλοι στη τελική ανάλυση ε, την αλήθεια την έχουν και οι Αμερικανοί, γιατί αλλιώ δεν θα είχαν συμμετάσχει μέχρι τώρα. Εγώ πιστεύω ότι οι δικοί μας στρατιώτες είναι πρόθυμοι να αγωνιστούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις το έπραξαν, αναγκάστηκαν να το κάνουν, όπου το έκαναν το έκαναν καλά και μερικές φορές απέφυγαν τη συμμετοχή. Ε, στη δική μας την ε, υπηρεσία, την Επιτροπή Άμυνας, ε, τιμήσαμε δύο λοχαγούς που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. Στο Κωσυφοπέδιο έγινε αυτό που σας είπα, δηλαδή τι έγινε, ήταν ένας στρατός ήταν ε, Γερμανοί στρατιώτες που έπρεπε να επιβλέψουν ένα μοναστήρι και εμφανίστηκαν ξαφνικά ε, περίπου 2.000 διαδηλωτές ε, με βόμβες Μολότοφ και κανονικά θα έπρεπε κανείς να πυροβολήσει για να προχωρήσουν αυτοί οι διαδηλωτές προς τον φυλασσόμενο χώρο. Αυτοί λοιπόν οι δύο λοχαγοί αποφάσισαν ότι δεν θα πυροβολήσουν, θα εκενώσουν το μοναστήρι και μετά θα αφήσουν το μοναστήρι στον όχλο. Και πράγματι το μοναστήρι κάηκε ολοσχερός, οι άνθρωποι όμως, οι ε, μοναχοί σώθηκαν. Τι έκαναν οι στρατιώτες, οι ε, στρατιώτες αποσύρθηκαν για να μην υπάρξει κλιμάκωση και ε, θεωρήσαμε ότι αυτή ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση και εμείς παρασημοφορήσαμε κυρίως τη σωστή απόφαση. Εγώ πρέπει να σας πω, ε, δεν το ήξερα παλαιότερα αυτό το μοναστήρι, μετά από αρκετά χρόνια το επισκέφτηκα και πραγματικά ε, εξοργίστηκα που το έκαψαν ο Γερμανός όμως αξιωματικός μου εξήγησε ότι εκείνο που κάηκε ήταν το ξύλινο κομμάτι, το παράρτημα του μοναστηριού. Το άλλο που είχαν κατασκευάσει οι Τούρκοι, αυτό παρέμεινε άθικτο και μπορεί να ανασυσταθεί. Τέτοιου είδου λοιπόν αποφάσει βλέπετε καλούνται σήμερα να τι λάβουν ακόμα και λοχίε και το κάνουν πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ ότι ο γερμανικό στρατό είναι τέλειο, αλλά ο γερμανικό στρατό είναι τώρα σωστά εκπαιδευμένο και υπάρχουν άνθρωποι και στα κατώτατα κλιμάκια που είναι σε θέση να αναλάβουν ευθύνε. Όσον αφορά τώρα τους ναζί στο γερμανικό στρατό, προφανώ. ε, ναζί δεν μπορούν να ενταχθούν σε στρατό δημοκρατών. Γι' αυτό λοιπόν κάθε χρόνο περίπου 24 στρατιώτες απολύονται, απομακρύνονται από το γερμανικό στρατό γιατί δείχνουν αυτά τα σύμβολα εχθρικά προς το κράτος, γιατί τοποθετούνται με εκφράσεις που δεν κρίνονται δημοκρατικές και μόλις διαπιστωθούν αυτά τα, αυτές οι περιπτώσεις, σας λέω, αποπέμπονται αυτή η στρατευμένη από το στράτευμα. Η AFD εμένα δεν μου αρέσει ως κόμμα και σε πολλούς δεν αρέσει στη Γερμανία. Αλλά τι να κάνουμε. Η AFD εξελέγει στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και στη τελική ανάλυση υπάρχει το κόμμα αυτό και σε άλλα κοινοβούλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον βαθμό λοιπόν που η οπαδοί του ΑΕΦΔ δεν εμφανίζονται με σλόγγαν και σύμβολα των Ναζί. Εντάξει, στη Γερμανία ε, ανησυχούμε ε, για την περίπτωση AFD, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Στην περίπτωση αυτή το ίδιο ισχύει και για το γερμανικό στρατό. Όσον αφορά τώρα την κοινή εξωτερική πολιτική, αυτό δεν είναι το δικό μου θέμα, δική μου αρμοδιότητα, αλλά προφανώς εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και εγώ είμαι υπέρμαχος αυτής της ε, διαδικασίας. Δεν υπάρχει το πριν και το μετά, υπάρχει μια διαδικασία όπου το ένα είναι σε απόλυτη συνάρτηση από το άλλο. Παραδείγματο χάρη, θα το έλεγα ε, φιλοσοφικά, η κανονιστική δύναμη του πραγματικού. Ε, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι παραδείγματο χάρη εμείς ε, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε συγκεκριμένη πολιτική έναντι της Ρωσίας, άρα το να συζητάμε αυτά τα θέματα δεν έχει σημασία. Ε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι η γερμανική κυβέρνηση να χαράσει μια πολιτική και να συντάσσεται με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Από την άλλη βέβαια ισχύει το ότι ε, στην εξωτερική πολιτική πρέπει να υπάρχουν πιο πολλά κοινά στοιχεία. Σας λέω, είναι ένα ε, παιχνίδι ισορροπιών. Το ένα, η μία πλευρά είναι απόλυτη συνάρτηση της άλλης. Πρόεδρος, πριν όμως ε, δώσω το λόγο σε εσά, θα ήθελα να πω το εξής, να ρωτήσω, στον Ολλανδικό στρατό υπήρξαν στρατιώτες που να αποπέμφθηκαν για πολιτικούς λόγους. Δεν μιλάω για στρατηγούς, χάρη, που να συνταξιδοτήθηκαν πρόωρα, αλλά μιλάω για ε, ακραίους, απλούς ε, που να αποπέμπτηκαν και μετά να ήρθαν και να έκαναν καταγγελία σε εσάς. Ε, αυτό είναι ένα συμπληρωματικό ερώτημα. Ε, προσωπικά δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Κοιτάζω κατά συνάδελφο, όχι από ό,τι βλέπω. Τουλάχιστον δεν έχουν γίνει γνωστά σε εμά ε, τέτοιου είδου περιστατικά. Βέβαια υπάρχουν και ξεκάθαροι κανόνες ό,τι αφορά την ε, παραβατική συμπεριφορά στην οποία επιβάλλονται κυρώσεις. Όμως, ας πούμε, απόπεμψη από το στρατιωτικό σώμα έχουμε σε περίπτωση χρήση κάναβη, για παράδειγμα. Όμως, για πολιτικούς λόγους να έχει υπάρξει τέτοια απόλυση, δεν το έχουμε ακούσει. Να πω δύο λόγια για κάποια ερωτήματα που δεν έχουν επευθυνθεί σε μένα προσωπικά, αλλά θεωρώ ότι είναι ενδιαφέροντα. Πρώτα απ' όλα, για την εσωτερική διαχείριση, που δεν ε, ξέρω ακριβώς τον Ολλανδικό όρο, όταν υπάρχει μια τέτοια συνεργασία, πάντα θα ανακύπτει αυτό το ζήτημα και στην προετοιμασία, ε, στο πλαίσιο ειρηνευτικών αποστολών, για παράδειγμα, εγώ τι έχω επισκεφτεί για να δω ακριβώ οι ε, δικοί μα ένστολοι πώ αντιμετωπίζονται σε ό,τι αφορά τι δημοκρατικέ ε, και θεμελιώδει αξίε. Όταν είχα πάει με τον κύριο Μπάρτελ στο Μαλί, το είχαμε δει προσωπικά. Με τον συνάδελφο μετά θα πάμε στο Αφγανιστάν για να απευθυνθούμε ε, στις στρατιωτικές μας δυνάμεις και να δούμε εκεί πώς ε, αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα. Και στο Μαλί και αλλού έχω δει ότι υπάρχουν διάφορα καθεστώτα ανάλογα με τον στρατό για τον οποίο εργαζόμαστε όταν έχουμε μικτές δυνάμεις, ε, κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά μεταξύ Γερμανίας και Ολλανδίας ε, και Ολλανδίας και Βελγίου, είναι λογικό να υπάρξουν και συστήματα καταγγελιών ε, για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των ενστόλων και θα πρέπει να βασίζονται φυσικά στις δημοκρατικές αξίες. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτή η συζήτηση ε, για την εσωτερική διαχείριση μεταξύ αυτών των χωρών. Τώρα, για τη στρατιωτική δραστηριότητα εν καιρό ειρήνης. Πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε από, από τις περιόδους ειρήνης, γιατί όταν φτάσουμε σε εμπόλεμες περιόδους, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν η σωστή κατάρτιση, η σωστή ηγεσία και θα πρέπει να τίθεται στην μέσα διάταξη αυτό το ζήτημα. Και εγώ και ο κύριος Μπάρτελ το κάνουμε, γιατί καταρτίζουμε έκθεση που καταθέτουμε ενώπιον του Κοινοβουλίου. Και το καλό για τη θέση μου είναι ότι δεν χρειάζεται να περιμένω να μου, θέσουν ερώτημα, μπορώ να το θέσω μόνο μου στην μέσα διάταξη. Ja, Είπατε και εσείς ε, ότι κάθε χρόνο ε, υποβάλλετε μία αίτηση στο Κοινοβούλιο. Το είπατε αυτό. Δεν ξέρω, υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, παρακαλώ. Ο Κρίστιαν. Λοιπόν, θέλω να κάνω μία παρατήρηση και θέλω να πω το εξής να αναφερθώ σε κάτι που είπε ο κύριος Μπάρτελς. Ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι η υποεπιτροπή πρέπει να ασχολείται με τα θέματα του τρόπου της Innenverführung, όπως λέει στα γερμανικά, του τρόπου με τον οποίο κάθε χώρα έχει οργανώσει το δικό της στρατό. Γιατί, διότι πάρα πολλοί από εμάς το έχουν δει αυτό όταν έχουν συμμετάσχει σε διάφορες αποστολές, ότι σε αυτό το θέμα της ε, ατομικής ηθικής ευθύνης ε, που αναλαμβάνει ένας πολίτης, αυτό δεν μπορεί πολύ εύκολα να συσχετιστεί με το διεθνές δίκαιο. Το έχουμε δει αυτό σε ασύμετρες απειλές. Δηλαδή, οι στρατευμένοι βρέθηκαν μπροστά σε αποφάσεις οι οποίες δεν αιτιολογούνταν από το διεθνές δίκαιο. Ας πούμε, συγκεκριμένα, σήμερα ε, σε συγκρούσεις ε, στη μάχη πάνω, ακόμα και με ανήλικα άτομα. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά αποκτούν μια νέα διάσταση και όσον αφορά την κοινή οργάνωση στην Ευρώπη γίνεται αυτή η συζήτηση και πρέπει να γίνει το πώς μπορεί να υπάρξει κοινή οργάνωση στρατιωτικών δυνάμεων. Δεν θέλω να ε, το ε, παρεξηγήσετε, αλλά θέλω να ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Μπάρτελ ε, και τους προκατόχους του, γιατί θεωρώ ότι ακριβώς αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να αιτιολογήσουν το ότι σήμερα μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για το δικό μας τον γερμανικό στρατό που υπηρετεί και τον ΝΑΤΟ και τις ε, εξωτερικές ε, επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να προβάλλεται σήμερα αυτή η γερμανική διάσταση στα τεκτενόμενα στο στρατό. Ο πρόεδρος και αυτό που βρίσκω και εγώ ε, πολύ ενδιαφέρον είναι ποια δικαιώματα έχουν οι στρατιώτες και τι ρόλο μπορούν να παίξουν. Αυτό ετέθηκε στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και επικαλούνται τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως επίσης και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Και τάσσονται ανεπιφύλακτα υπέρ του ότι οι στρατιώτες και οι στρατευμένοι δεν χάνουν τα δικαιώματά τους με το που μπαίνουν στο στρατό. κατά άλλο παραμένουν πολίτες ενός συγκεκριμένου κράτους. Το Μαλί αναφέρεται ένα παράδειγμα. Εκεί έχουμε διαφορετικές αποστολές, διαφορετικές επιχειρήσεις, έχουμε ε, στρατευμένους από διάφορα κράτη που βρίσκονται στο Μαλί. Το ένα είναι εκπαιδευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άλλο λέγεται Μινούσμα, ε, εκεί συμμετέχουν και τα Ηνωμένα Έθνη. Και μετά έχουμε και τους Γάλλους φίλους που έχουν σε διμέρες επίπεδο την αποστολή Μπεκά ε, ως εκ τούτου, ως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι μεν έχουμε μία πολιτική έναντι του Μαλή, αλλά έχουμε και διαφορετικά νομικά πλαίσια ε, που ισχύουν. Άρα δηλαδή πώς θα τα συνδυάσουμε αυτά μακροπρόθεσμα. Είπε εσύ προηγουμένω ω παράδειγμα, ο στρατιώτη έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του έναν, ε, ένα παιδί, έναν ανήλικα. και μπορώ να φανταστώ ότι οι Γάλλοι κυρίως προσπαθούν να εξολοθρεύσουν, θα το πω όπως είναι πραγματικά αυτές τις εστίες και ξέρετε τι κάνουν εκεί, δεν κοιτάνε αν είναι ανήλικας αυτός που πέταξε τη χειροβομβίδα ή όχι, ε, ούτε καν ε, θέτουν το θέμα νομικά ότι αν δηλαδή αιτιολογούνται όλα αυτά ε, τα οποία διαδραματίζονται στο βορρά, όπου οι στρατιώτες ε, ε, χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν ένα στρατό ή ναι, όχι. Αυτά εμφανίζονται στην κοινή γνώμη και ξαφνικά προκύπτει ένα τελείως διαφορετικό νομικό πλαίσιο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εσείς ε, με τους συναδέλφους σας σε ευρωπαϊκό επίπεδο συζητάτε, υπάρχουν ε, τέτοιου είδου συναντήσει ε, φόρα όπου να τα συζητείτε όλα αυτά ή τα αφήνετε έτσι να τρέχουν και να λέτε, και λέτε εντάξει αν κάνουμε άλλη εσωτερική διαχείριση του ενός κράτους και άλλη ε, σε άλλες χώρες. Και στην Γερμανία ας πούμε ισχύει το τεκμήριο τη αθότητα Στη Γαλλία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην ισχύει. Τι κάνετε, λέτε εντάξει δεν πειράζει, έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Εγώ πιστεύω ότι όταν συνεργάζεται κανείς και ακολουθεί μία συγκεκριμένη πολιτική, τότε θα πρέπει να ισχύουν καταστάσεις όπου για τους ε, στρατευμένους, ε, τους Ευρωπαίους, ισχύουν παντού τα ίδια. Τι γνώμη έχετε? θεωρώ ότι αν δείτε στο Μαλί τι γίνεται, βλέπετε ότι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Πήγαμε μαζί. Πέραν των Γάλλων έχουμε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ Ολλανδίας και Γερμανίας και μετά υπάρχουν 12 άλλες ε, στρατιωτικές δυνάμεις. Αν δείτε ε, τις διαδικασίες που ακολουθούνται, τα πρότυπα ασφαλείας και ούτε καθεξής, σίγουρα δεν έχουμε σκεφτεί εκ των προτέρων πώς μπορούν να λυθούν τυχόν προβλήματα. Και μπορεί να είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ε, τι γίνεται όταν έχουμε αξιωματικούς από διαφορετικές χώρες που εμπλέκονται σε μια κοινή επιχείρηση. Από τη μία πρέπει να υπάρχει κάποια ανταπόκριση, από την άλλη να μην είναι υπερβολική, να είναι σωστή. πριν από δύο εβδομάδες όταν ήμασταν στην Νότια Αφρική μαζί με κάποιους ε, συναδέλφους ε, τα εξετάσαμε τα πράγματα και είπαμε ότι ως ενίγορο των βετεράνων μαζί ε, με τη Γερμανία, την Νορβηγία και άλλους που θα συμμετάσχουν να υπάρχει ανταλλαγή μεταξύ μας για τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στο έργο μας για να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα προς το συλλογικό. Και το ψήφισμα αυτό που θα την επόμενη φορά σίγουρα Τώρα που προσυπογράφονται από μία σειρά συνηγόρου σε διάφορε χώρες, για μας είναι το πρώτο βήμα συνεργασία. Και στη συνέχεια μπορεί να αποτελέσει υλικό για εσάς, για να δείτε τι βήματα μπορούν να γίνουν και τι πλαίσια μπορούν να δημιουργηθούν. Υπάρχουν λοιπόν δεσμοί συνεργασία. Και νομίζω ότι ήταν και από τις πρώτες, τους πρώτους που ε, εμείς δηλαδή που πήγαμε σε κοινέ αποστολές και ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας και παράδειγμα προς για άλλους. Δεν ξέρω αν ε, τα κατάλαβα καλά, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια οργάνωση που συναντιέται μία φορά το χρόνο, ΑΜΚΟΑΦ, είναι ένας ε, οργανισμός ε, στον οποίο εκπροσωπούνται πάρα πολλοί συνήγοροι από ολόκληρο τον κόσμο. Φέτος εκπροσωπήθηκαν 130 οργανώσεις αυτών των διεθνών οργανισμών, εκ των οποίων 20 περίπου ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Και μπορούμε το ψήφισμά μας, αν θέλετε, να σας το διαθέσουμε. Έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα, το πώς μπορεί κανείς ε, να ε, κοινοποιεί τα δικαιώματα περί ε, προσφυγής στο συνήγορο. Μετά υπάρχουν τα δικαιώματα των στρατευμένων. Και αν δούμε την περίπτωση του Μαλή, εκεί το βασικό ερώτημα είναι ποιος ηγείται, ποιος καθοδηγεί τις ε, στρατιωτικές ε, δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο Μαλί. Τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα από ό,τι είπατε. Έχουμε Γερμανούς, Συμβουλευτική Επιτροπή, έξι Γερμανούς που ε, παρουσιάζουν, καθοδηγούν για διάφορα προγράμματα εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτοί αποσπώνται ε, για τρία χρόνια, ε, γνωρίζουν ε, πάρα πολύ καλά τα όλα θέματα και τα καταφέρνουν μια χαρά. Μετά, πέρα από τους Γερμανούς, έχουμε την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 500 στρατευμένοι, περίπου 145 Γερμανοί. Από τους 145, οι 7 είναι εκπαιδευτές αλλά 145 πάλι οι Γερμανοί. Τεράστια δαπάνη. Τώρα κατά πόσον αυτό είναι αποτελεσματικό δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος. Ε, κατά τα άλλα η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται ότι εμείς είμαστε οι μόνοι που κάνουμε εκπαιδευτή. Τι λέτε, οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, οι Αμερικανοί, όλοι αυτοί εκπαιδεύουν και οι Γάλλοι ενδεχομένως σε διμερές επίπεδο, οι ειδικέ δυνάμεις και αυτοί. Άρα δηλαδή παντελής έλλειψη συντονισμού. Έχουμε την αποστολή των ε, Ηνωμένων Εθνών που εκεί συμμετέχουν αρκετοί Ευρωπαίοι, Γερμανοί, Ολλανδοί, Σουηδοί, από πάρα πολλές ε, εθνικότητες που συμμετέχουν και αυτοί σε αυτές τις επιχειρήσεις, κατ' ουσίαν θα έπρεπε να υπάρχει συντονισμός για όλα, για τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, εθνικές ε, αντιπροσωπείες. Αυτό υπήρξε στα Βαλκάνια, δηλαδή όταν τα πράγματα επιδεινώθηκαν στα Βαλκάνια, εκεί υπήρξε απόλυτο συντονισμός. Υπήρχε ένας επίτροπος των Ηνωμένων Εθνών για την Βοσνία Ερσεγοβίνη, ο οποίος μπορούσε να ακυρώσει αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν έκρινε ότι ε, δεν ήταν καλές. Μετά στείλαμε ε, δήμαρχο στο Μόσταρ ε, για να είναι πραγματικός δήμαρχος, όχι απλά για να συζητάμε τους πολίτες. Στα Βαλκάνια δηλαδή για ένα κάποιο χρονικό διάστημα πράγματι υπήρξε μια ουσιαστική οργάνωση γιατί ήταν απολύτως απαραίτητο. Στο Αφγανιστάν δεν το καταφέραμε ποτέ. Ε, πολλές δραστηριότητες παράλληλες στο Αφγανιστάν Αμερικανών, του ΝΑΤΟ, ε, των Αφγανών. Και στο Μαλί τα ίδια. Μόνο που στο Μαλί δεν έχουμε Αμερικανούς. Ως εκ τούτου, αν δεν λάβουν οι Ευρωπαίοι τα πράγματα στα χέρια τους και δεν μπουν ότι οι Γερμανοί και οι Γάλλοι κάπως πρέπει να τα βρούνε, τότε θα είναι πάρα πολύ κρίμα. Θα μπορούσε, παραδείγματο χάρη, ο εκπρόσωπο ε, των ΗΠΑ να συντονίζει την κατάσταση. Στο Μαλί αυτή τη στιγμή, και καλό είναι αυτό, δέχεται πολύ μεγάλη βοήθεια από πολλά κράτη που στέλνουν στρατευμένους, όχι όπως παλαιότερα και τώρα στο Αφγανιστάν. Στο Μαλί υπάρχει επαρκής ε, ε, βοήθεια σε διμερές επίπεδο και μη στρατιωτική βοήθεια, αλλά σας λέω, παράλληλες ε, δομές. Βέβαια, η κυβέρνηση του Μαλίτα τα δέχεται όλα, αλλά μην φανταστείτε ότι η κυβέρνηση είναι σε θέση να τα συντονίσει, γιατί αν ήταν σε θέση να τα συντονίσει, συντονίσει δεν θα ήταν και αυτοί παρόντες. Νομίζω ως εκ τούτου ότι είναι ένα αίτημα που πρέπει να εκφραστεί, να υπάρχει καλύτερο συντονισμός, καλύτερη καθοδήγηση, γιατί σας λέω και πάλι στα Βαλκάνια τα καταφέραμε. Κακό παράδειγμα, είχαμε έναν Γερμανό εκπρόσωπο των ΗΕ στο Αφγανιστάν, έμεινε εκεί δύο χρόνια, έγραψε ένα βιβλίο και αν διαβάσει κανείς το βιβλίο θα ε, δει πόσο αδύναμος ήταν αυτός ο Γερμανός στο Αφγανιστάν, γιατί δεν του επιτρεπόταν τίποτα. Ως εκ τούτου ε, θα πρέπει να μεταφέρουμε όχι μόνο τα μέσα, αλλά και την αποφασιστικότητα και ε, η αποφασιστικότητα όσον αφορά την αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν νομίζω ότι ταιριάζουν αυτά τα δύο πράγματα και αυτό είναι πολύ απογοητευτικό για τους στρατευμένους. Πρόεδρος, πολύ ωραία. Αν ε, δεν θέλει κανείς να λάβει το λόγο, ευχαριστώ πολύ τους ε, δύο προσκεκλημένους και θα έλεγα αυτά όλα που μας είπατε να τα σκεφτούμε, να τα επεξεργαστούμε όχι μόνο σε σχέση με το μαλλί αλλά και με την αναγκαιότητα να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα των ε, στρατευμένων τόσο στις ε, πατρίδες τους, αλλά και όταν βρίσκονται σε εξωτερικές αποστολές. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Ευχαριστώ και τους αδέλφους που πέρασαν από εδώ και παρακολούθησαν. Στις, ε, στη μία η ώρα έχουμε την ομάδα Κάγκουρου και σας είπα, αν θέλετε μπορούμε εκεί να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Κατά τα άλλα, ε, αν όχι, εύχομαι σε όλους όσοι συμμετείχαν Καλή όρεξη. Ε, θα συνεχίσουμε στις 2.30 το απόγευμα. Γεια σας.